Friends, colleagues, can I Παρακαλώ να καθίσετε συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση αυτή που προκαλεί αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον λόγω θέματος προστασία δεδομένων στην διατλαντική αυτή προοπτική. Το πρόγραμμα λέγει ότι κανονικά θα κηρύξει την έναρξη ο Φερνάντο Λόπες Αγουιλάρ, δηλαδή όχι εγώ. Έχω την τιμή να προεδρεύσω τη συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα. Έχουμε εδώ ε, μια πλειάδα εξαιρετικών εμπειρογνωμόνων ομιλητών και θα αναφερθούν σε ε, πολλά θέματα και θα καλύψουν ε, ε, νομίζω το ενδιαφέρον. Σας έχω τον εισηγητή εδώ, τον κύριο Ιάν Φίλιπ Αλμπρεχτ από τους Πρασίνους, Γερμανός. Κάντε παρακαλώ μια σύντομη εισαγωγή κυρία Άλμπρεχτ και μετά θα περάσουμε στους ομιλητές του πάνελ και θα ακολουθήσουν ερωταπαντήσεις. Κύριε Άλμπρεχτ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εισήγηση, την εισαγωγή. Βλέπω τώρα με χαρά μου ότι εσείς προεδρεύετε τη συνεδρία σας. Θα προσπαθήσω να είμαι ως το δυνατόν πιο σύντομος στα λόγια που θα σας απευθύνω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τα τελευταία χρόνια πολλές φορές ε, διατυπώσει το αίτημα για μια συνολική ε, δέσμη προδιαγραφών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε θέματα συνεργασίας με τρίτα κράτη, ιδιαίτερος βέβαια με τους ε, εταίρους με τους οποίους έχει πιο στενή συνεργασία, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συχνά λοιπόν έχουμε διατυπώσει το αίτημα για μια συμφωνία πλαίσιο τώρα, χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Το αίτημα αυτό καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό, γιατί αναμεινόμαστε ακόμη περισσότερο σε θέματα αστυνομίας, αστυνομικής συνεργασίας και δικαστική συνεργασία και τον προσδιορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών ε, με βάση τον ε, χάρτη των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Έτσι, πέραν του καθημερινού έργου που έχει να κάνει με την συζήτηση συμφωνιών σχετικών με την προστασία των ε, τραπεζικών δεδομένων και άλλων που επεξεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ, ε, επεξεργαζόμαστε και μια σειρά βασικών αρχών, δηλαδή κοινών προδιαγραφών στις οποίες αποσκοπούμε να καταλήξουμε όταν θα υπάρχει περισσότερη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια διαπραγματευτική εντολή και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε από τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Εμείς από πλευράς μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ε, συζήτηση αυτή θέλουμε να ε, βοηθήσουμε έτσι ώστε να καταλήξουμε το ταχύτερο δυνατό σε μια πιθανή συμφωνία και να ε, εμπλακούμε σε μια συζήτηση η οποία θα αφορά όχι μόνο τη συγκεκριμένη αυτή συμφωνία αλλά η οποία μακροπρόθεσμα θα ε, μας επιτρέψει να διατυπώσουμε τις δικές μας προδιαγραφές με την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν που έχουμε σήμερα και με την παρουσία ε, υψηλών προσκεκλημένων για ανταλλαγή απόψεων, για διαμόρφωση ιδεών ως προς το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει, τι μορφή και περιεχόμενο θα πρέπει να έχει αυτή η συμφωνία, μια τέτοια συμφωνία. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το να έχουμε εδώ στην αίθουσά μας και τους ευρωβουλευτές, έτσι ώστε και αυτοί να εμπλακούν στη συζήτηση και να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Για αντίστοιχη ακρόαση που οργάνωσα εγώ ίδιος, είχα την ευκαιρία να μιλήσω πριν από μερικούς μήνες αποτέλεσε και αυτή μια πολύ ενδιαφέρουσα εκκίνηση με διαφορετικές προοπτικές και κόμματα που ακούστηκαν. Διαφορετικές πλευρές και οπτικές γωνίες δηλαδή εκφράστηκαν. Και ελπίζω ότι και η σημερινή ακρόαση θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τη γραμματεία της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών, η οποία έχει σκληρά εργαστεί για την οργάνωση της παρούσας ακρόασης. Καλώς ήρθατε όλοι και περιμένω με χαρά να ακούσω τις ε, ομιλίες σας. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Και παρακαλώ τώρα τους ομιλητές. Θα ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Προεδρία, μετά της Ένωσης και βέβαια και τους ε, φίλους από την άλλη πλευρά της, ε, του κτηρίου, της αίθουσας. Το ενδιαφέρον ότι είχαμε διατλαντική συνεργασία ε, επί έτη πολλά για την ασφάλεια. Τώρα γυρίζει κάπως ο τροχός και έχουμε διατλαντική συμφωνία, συνεργασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα παρακαλέσω λοιπόν πρώτα την κυρία Φρανσουάζ Λεμπάγη, Γενική Διευθύντρια τη Γενική Διευθύνσεω Δικαιοσύνη για θέματα δικαιοσύνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά θα ακούσουμε τον κύριο Στεφάν Ντεκλέρκ, Υπουργό Δικαιοσύνη του Βελγίου, άρα προεδρεύοντα και εκπρόσωπο τη Προεδρία του Συμβουλίου. Και στη συνέχεια τον κύριο Κέναρτ, πρεσβευτή στην αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις τους και μετά θα έχουμε ένα χρονικό περιθώριο για ερώτα αποκρίσεις. Παρακαλώ, κυρία Λεμπάλια. Ευχαριστώ την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών που πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή την ακρόαση σήμερα. Όχι μόνο είναι καλή η πρωτοβουλία αυτή, αλλά είναι και εύθετη χρονικά. Όταν συζητάμε το θέμα της συμφωνίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το τι μοιραζόμαστε με τις Ηνωμένε Πολιτείες και να σταθούμε στη μακρά συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Η συνεργασία αυτή γίνεται επί τη βάση των αρχών μας για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και γενικότερα τις κοινέ αξίες. Νομίζω ότι η αμοιβαία πληροφόρηση σε τομείς όπου υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον θα βοηθήσει και την καταπολέμηση του εγκλήματος και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτού του είδους η εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας όχι μόνο είναι σημαντική αλλά θα τη χαρακτήριζα απαραίτητη. Η συνεργασία μας έχει σαν στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, των οικονομικών δομών στήριξης της τρομοκρατίας και της ανταλλαγής γνώσεων γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Συνεργαζόμαστε στενά λοιπόν με τη ΣΥΠΑ όπως γνωρίζετε έχουμε πολλά διατλαντικά μέσα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί η δημιουργία τους και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μηχανισμών διευκόλυνσης της ομαλής ανταλλαγής πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων για στοχευμένους κάθε φορά χώρους. Ξέρετε για τα PNR, τα TFTP κτλ. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών υπάρχει ένα μοσαϊκό εδώ συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Αυτές οι δυνατότητες όλοι μας συμφωνούμε ότι είναι αρκετά χρήσιμες. Το αποτέλεσμα δεν είναι βέβαια πάντα ικανοποιητικό ακριβώς λόγω αυτής της φύσεως του μοσαϊκού που χαρακτήρισα. Αλλά ε, παρόλα αυτά βλέπουμε το θέμα της προστασίας των πολιτικών δεδομένων σαν θεμελιώδες ε, ε, θα έλεγα δικαίωμα δείχνουμε αποφασιστικότητα για να διορθώσουμε κάπως την κατάσταση, να την καταστήσουμε πιο ικανοποιητική. Η ανταλλαγή ε, πληροφοριών είναι κρίσιμη για τα θέματα της εθνικής ασφάλειας ε, και της υπηρεσίες καταστολής, αλλά δεν θεωρούμε ότι η ασφάλεια ε, και η προστασία των ιδιωτικών στοιχείων είναι δύο αντιφατικά χαρακτηριστικά και αυτά είναι τα θεμέλια αν θέλετε της αντίληψης η οποία κυριαρχεί πίσω από τις προτάσεις τις οποίες μέχρι τώρα έχουμε κάνει. Απαιτείται να ενισχύσουμε και την δικαστική συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και την ανταλλαγή δηλαδή στον τομέα αυτό των απαραίτητων δεδομένων και να το κάνουμε αυτό χωρίς να ξεχάσουμε την σημασία που έχει ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι σαφές ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάτι το οποίο θα έλεγα έχει αντιμετωπιστεί με αντιφατικό τρόπο, έχει προκαλέσει πάρα πολλές διαφωνίες και έχει συζητηθεί επανειλημμένα το θέμα της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εμείς θα θέλαμε στα πλαίσια της συνεργασίας και των συμφωνιών μας με τη ΣΥΠΑ να επιλύσουμε τα θέματα αυτά επί τη βάση ακριβώς των αξιών των κοινών στις οποίες προαναφέρθηκα. Πέραν των κοινών αυτών αξιών έχουμε και συστήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και, και του ιδιωτικού χαρακτήρα των προσωπικών στοιχείων που δεν είναι ταυτόσιμα. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξομαλύνουμε τα δύο συστήματα αυτά προστασίας, ε, να τα καταστήσουμε ομοιογενή και αυτό θα προωθήσει την νομική βεβαιότητα και ασφάλεια και προστασία των πολιτών μας. Τα συστήματα, όπως είπα, ε, προστασίας δεδομένων δεν είναι α, ταυτόσιμα, αλλά έχουμε και διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την συλλογή των προσωπικών δεδομένων και την αμοιβαία χρήση των δεδομένων αυτών και αυτό έχει σημασία για την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων αυτών ή της εποπτείας ε, του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων αυτών από τις αρμόδιες αρχές. Οι διαφορετικές αυτές ε, αντιλήψεις λοιπόν κάνουν την κατάσταση πάρα πολύ περίπλοκη έτσι ώστε να καταλήξουμε σε αμοιβαία αποδεκτά επίπεδα προστασίας δεδομένων. Στην Ευρώπη, όπως έχω ήδη πει, μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο βάρος, γιατί τα προσωπικά δεδομένα είναι πλέον, θεωρούνται πλέον ένα, ένα ουσιαστικό δικαίωμα, ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Η πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για τις κατευθυντήριες διαπραγματευτικές γραμμές στα πλαίσια της επικοινωνίας μας με τους Αμερικανούς ομολόγους είναι ήδη γνωστές. Έχουμε τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να διασφαλίσουμε ένα υψηλότατο επίπεδο προστασίας στην περίπτωση μεταφοράς προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι ε, συμβατό και με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Φυσικά δεύτερος στόχος είναι να αποκαταστήσουμε ένα απλό, συνεκτικό, νομικά δεσμευτικό και απαραβίαστο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτή η βασική αρχή του ενιαίου και συνεκτικού επίπεδου προστασίας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το σύνολο των διαπραγματεύσεων. Και ο τρίτος στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα έχει σαν στόχο την ουσιαστική εφαρμογή μια σταθερής βάσης συνεργασίας ανάμεσα στην Ένωση από τη μία και τη ΣΥΠΑ από την άλλη. Συμπερασματικά λοιπόν στόχος μας σε αυτή τη φάση είναι η απαραίτητη σε υψηλό επίπεδο προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν συγκεκριμένες ε, υποχρεώσεις αυτών που ελέγχουν τα δεδομένα και τους στόχους για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα αυτά, όπως επίσης και ελέγχουν τον πλήρη σεβασμό των, επιπέ... των συμπεφωνημένων επιπέδων προστασίας. περιμένουμε να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες απλουστευμένες μορφές δεδομένων που θα ε, πρέπει να εφαρμοστούν ε, με ενιαίο τρόπο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στα ποινικά θέματα. Αυτά όλα λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία που οδηγούν σε αυτό που ονομάζουμε νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Βασικά λοιπόν καθορίζουμε ένα κατάλογο αρχών που θα εφαρμόζονται σε όλες και θα περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα στην Ένωση και τη ΣΥΠΑ και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη της Ένωσης και τη ΣΥΠΑ έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αναγνώριση του απαραβίαστου των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι δύσκολη η προσπάθεια αυτή, δεν υποτιμούμε το βαθμό δυσκολίας, αλλά είναι κάτι το απαραίτητο εφόσον θέλουμε να καταργήσουμε τα εμπόδια στις διατλαντικές αυτές σχέσεις και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Ένωση, ένα σύστημα το οποίο ταυτόχρονα θα ενισχύει τα επίπεδα ασφαλείας και θα ενισχύει επίσης και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη. Ευχαριστώ. Ξέχασα να πω πως ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή η συνάντηση έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διοικητικό επίπεδο έχει ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με τη ΣΥΠΑ εδώ και χρόνια και το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε δημόσιος διάλογος, δεν υπήρχε πολιτική εποπτεία των διαπραγματεύσεων αυτών που αφορούσαν τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει χώρος για ένα σωστό δημοκρατικό ανοιχτό διάλογο. Ο κύριος Ντεκλέρκ λοιπόν εκ μέρου της Βελγικής Προεδρίας, της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ολλανδικά γιατί μου είπαν ότι μπορώ, λέει ο Υπουργός Ντεκλέρκ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα εκ μέρους της ε, Προεδρίας, της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Και παρακολούθησα και τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το SWIFT. Τώρα συνεχίζουμε τη συζήτηση, προχωράμε ακόμα περισσότερο για τη συμφωνία πλαίσιο που πρέπει να διαπραγματευτούμε. Είναι προφανές λοιπόν ότι η προστασία δεδομένων είναι πολύ σημαντική για όλους, για όλες τις χώρες και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι θεμελιώδη ζήτημα. Και πολιτικά έχει μεγάλη σημασία, αλλά και γενικότερα πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητα και αποτελεί προτεραιότητα της Βελγικής Προεδρίας. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε γρήγορση όσον αφορά το θέμα της προστασίας δεδομένων. Είναι προφανέ λοιπόν για την Προεδρία μα ότι κάθε πρωτοβουλία σχετική με αυτό το θέμα τη στηρίζουμε για την προστασία δηλαδή των προσωπικών δεδομένων και στα πλαίσια διατλαντικών συμφωνιών και για το επίπεδο στο οποίο μπορούμε να αποφασίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσπαθούμε λοιπόν να ενισχύσουμε ό,τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για διαπραγματεύσεις στον τομέα αυτό και να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Το κείμενο το οποίο έχει προχωρήσει έχει μελετηθεί δύο φορές στην ομάδα εργασίας Stadex, δύο φορές στα πλαίσια της Επιτροπής Συντονισμού ΚΑΤΣ και είναι και στην ημερήσια διάταξη ε, αργότερα σήμερα πάλι σε συνεδρίαση της ΚΑΤΣ για να συζητηθούν παρετέρω τα τεχνικά στοιχεία όσον αφορά αυτό το θέμα. Φιλοδοξία μας λοιπόν είναι την ε, εντολή του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου να την ε, φέρουμε σε πέρας. Και ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε σε αυτό. Τώρα, Εξαιτία ε, τη ρύθμιση που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να δοθούν μόνο εφόσον αυτοί που τα ζητάνε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο προστασίας. Πρόκειται για το, τη Συμφωνία 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για άλλες ρυθμίσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2008 κάθετος 977 απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια υπάρχουν εντάσεις για το θέμα αυτό ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η Αμερικανική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων που είναι από το 1977, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, έτσι λοιπόν, δεν προστατεύουν βάσει αυτής της νομοθεσίας τα δεδομένα που αφορούν Ευρωπαίους πολίτες. Για 10 χρόνια λοιπόν προσπαθήσαμε να βρούμε τις κατάλληλες ε, εγγύησεις έτσι ώστε να προστατεύονται και οι Ευρωπαίοι πολίτες και διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια τέτοια συμφωνία. Εδώ και 10 χρόνια λοιπόν έχουν υπάρξει τομεικές συμφωνίες, ειδικέ ρυθμίσεις, που είναι όμως διαφορετικές για κάθε τομέα και έτσι υπάρχουν διαφορές που έχουν σαν αποτέλεσμα να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παζλ. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο οι υπάλληλοι, οι αστυνομικοί και λοιπά να μπορούν να μας καλύψουν όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, περιπλέκεται και για τους πολίτες το θέμα. Γιατί ένας πολίτης τελικά δεν ξέρει με ποιο τρόπο προστατεύονται τα προσωπικά του δεδομένα ή με ποιο τρόπο εκτίθεται. Έτσι λοιπόν, για διαφορετικά δεδομένα έχουμε διαφορετικές συμφωνίες, για διαφορετικού είδους δεδομένα. Για να μπορεί να υπάρχει μια ανταλλαγή δεδομένων, που να προστατεύεται όμως από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το κάναμε αυτό όσον αφορά το PNR και για το SWIFT. Έχουμε δηλαδή πρόσφατα σχετικές πολιτικές εμπειρίες. Το γενικό πλαίσιο ρύθμισης πάντως για την προστασία των δεδομένων θέλουμε να υπάρχει και γενικά και όχι μόνο ανατομέα. Έτσι ώστε στο μέλλον να μην χρειαστεί πάλι και ξανά ανατομέα να συμφωνούμε κατά περίπτωση. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε την κατεύθυνση αυτή που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει εξάλλου να είμαστε και ρεαλιστές. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να ξέρουμε ότι μια γενική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για προστασία δεδομένων ποτέ δεν θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και τα πάντα. Πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες θα πετούν μια ειδική συμφωνία για το συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, δεδομένα τα οποία ε, διατηρούμε δεν μπορούν να, δεν είναι δυνατόν να εμπίπτουν σε ένα και μόνο πλαίσιο. Το γεγονός δε ότι σύντομα και μάλιστα μετά από έτοιμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα υπάρξουν νέε διαπραγματεύσει με τι Ηνωμένε Πολιτείε ε, για το PNR. Είναι κάτι το οποίο δείχνει ακριβώς ότι μια γενική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων δεν αποκλεί να υπάρχουν και κατατομέα συμφωνίες. Η συμφωνία πλαίσιο λοιπόν αποτελεί αν θέλετε, μια ομπρέλα, μια, ένα γενικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων, αλλά δεν ε, καλύπτει πλήρως, διότι υπάρχουν κενά τα οποία θα καλύπτονται με ειδικέ συμφωνίες ανατομέα, για ειδικέ περιπτώσεις, για ειδικέ αρχές και ειδικά μέτρα προστασίας εφόσον χρειάζεται. και αν μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι, είναι μια χώρα η οποία απαιτεί την ίδια προστασία δεδομένων. Πρέπει, όντως, να μπορούμε να εγγυθούμε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο προστασίας. Άρα να ισχύει η προστασία αυτή και για τους Ευρωπαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Ευρώπη. Στο, στη Συμφωνία 108 λοιπόν του Συμβουλίου της ε, Ευρώπης αναφέρεται όπως επίσης και στα πλαίσια της οδηγίας του 2008 ότι τα δεδομένα συλλέγονται για έναν σαφή και συγκεκριμένο λόγο και σκοπό. Για παράδειγμα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για ανεξάρτητους στόχους. Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται κατά με το στόχο και όχι κατά υπερβολή δεν πρέπει να συλλέγονται περισσότερα στοιχεία από όσα χρειάζονται για το συγκεκριμένο στόχο. Για το συγκεκριμένο στόχο. Και οι πολίτες πρέπει να μπορούν να ενημερωθούν σχετικά. Ένας πολίτης πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Ένας πολίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει, αν υπάρχει κάποιο λάθος δηλαδή, να το διορθώσει στα προσωπικά του δεδομένα. Επίσης ο πολίτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να προσφύγει σε αρχές για την προστασία των δεδομένων. Τον Οκτώβριο του 2009, ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το High Level Data Protection Group, για τρία χρόνια δούλεψε και κατέληξε σε γενικές αρχές της συμφωνίας. Οι αρχές αυτές είναι αρχές αυτές οι οποίες αποτελούν και τη βάση για τις συνομιλίες που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. το επίπεδο προστασίας. Είναι μια έννοια που πρέπει να είναι σαφής. Πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε. Το δικαίωμα ενός ε, ατόμου είναι να μπορεί να προστατευτεί σε υψηλό επίπεδο και να μπορούμε να εγγυθούμε την προστασία αυτή χωρίς να υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν διαφορετικά δικαστικά συστήματα, οπότε το κάθε σύστημα βέβαια διαφέρει, αλλά η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να θέσει το πλαίσιο. Το να υπάρχουν διαφορές δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό που έχει σημασία είναι και ο Ευρωπαίος πολίτης και ο Αμερικανός πολίτης να έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία να καθορίζονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να είναι κάτι συγκεκριμένο. Και ακριβώς αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται και οι διαβουλεύσεις που έχουμε. Όπως συμβαίνει και με άλλες οδηγίες, όντως οι οδηγίες εφαρμόζονται μερικές φορές διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, το ίδιο περίπου ισχύει και σε αυτή την περίπτωση στη συμφωνία αυτή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μία δομή που να λειτουργεί καλά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίσει να μπορούμε να συνεργαζόμαστε καλά η Ευρώπη με τις Ηνωμένε Πολιτείε, δίνοντας την κατάλληλη προστασία στους πολίτες μας. Έχουμε δουλειά ακόμα. Έχουμε τις αρχές, αλλά πρέπει να τις κάνουμε συγκεκριμένες και πρέπει να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ελπίζουμε μέσα στην εντολή αυτή το Δεκέμβριο δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε προχωρήσει στην πολιτική συζήτηση, σε συζήτηση δηλαδή που προβλέπεται στο Συμβούλιο με τα 27 κράτη-μέλη. Βέβαια η εντολή αυτή έδινε τις βάσεις για συνομιλίε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε επαφές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά και μετά. Η Προεδρία θα φροντίσει με την Επιτροπή να προχωρήσει στις συνομιλίες και η Επιτροπή θα ενημερώνει για το επίπεδο των ε, συνομιλιών, πώς έχουν προχωρήσει. Σίγουρα η Επιτροπή θα ενημερώσει και το Κοινοβούλιο, το οποίο θα είναι πάντα ενημερωμένο. Είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μας. Πιστεύουμε ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι θέσεις μας και να τολμήσουμε να προχωρήσουμε σε ένα διάλογο ο οποίος να μην μας ε, εμποδίσει να προχωρήσουμε, να μην νιώθουμε καμία απειλή. Πρέπει να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Και είμαι πεπισμένος ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν ένα στόχο που και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή και για το Συμβούλιο είναι κάτι πολύ σημαντικό και έτσι μαζί θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βρούμε μια λύση. Επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα, πριν από το Δεκέμβριο, πριν φτάσουμε στις συνομιλίες ε, του Δεκεμβρίου, που μου δίσατε την ευκαιρία, κυρία Πρόεδρε, να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε εδώ και να συμμετάσχετε στη συζήτηση αυτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πράγματι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στο διάλογο, αλλά και στην ψηφοφορία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Επόμενος ομιλητής είναι ο πρέσβης Κινάρτ από την ε, αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπετε ακόμα κι αν επίσημα θα έχουμε διαπραγματεύσεις που διακυδεύονται και εθνικά συμφέροντα, πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πάνω σε μια μερίσια διάταξη που έχει να κάνει με την ασφάλεια και με τις κοινωνικές μας αξίες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ κυρία Ινετφέλτ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άλμπρεχτ για την έκθεση και όλα τα μέλη της Επιτροπής και τους εδώ παρισταμένους. Είχα αρκετέ φορέ την ευκαιρία να απευθύνω το λόγο, δηλώνοντα σε εσά, δηλώνοντα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε αναγνωρίζουν και σέβονται το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιθυμούμε την εμβάθυνση των σχέσεών μα με το Κοινοβούλιο σα. Σε αυτό το στόχο αγωνιζόμαστε. Και πρόκειται για ένα μήνυμα το οποίο δεν απευθύνω μόνο εγώ εδώ ω πρεσβευτή των ΗΠΑ, αλλά και ο αντιπρόεδρο Βάιντεν, τον έχει, το έχει πράξει και η υπουργό των Εξωτερικών, κυρία Κλίντον, και ο κύριος Πολετάνο και πολλοί άλλοι ε, αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ που έχουν επισκεφθεί το κοινοβούλιο σας ε, το τελευταίο διάστημα. Και νομίζω ότι αποτελεί αυτό και σαφή ένδειξη του σεβασμού που τρέφει ο πρόεδρος Ομπάμα για το κοινοβουλίο σας. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να αναφερθώ σε ορισμένους τομείς. Ένας είναι οι κοινέ μας αξίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων, του ιδιωτικού βίου, τις κοινέ μας εργασίες, το κοινό μας έργο στο θέμα αυτό, τις ε, ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς ως κυβέρνηση στην εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία και επίσης το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην κοινή μας συνεργασία. Κοινέ αξίες καταρχάς. Και εν μέρει αναφέρθηκε αυτό νωρίτερα. Έχουμε κοινέ αξίε κοινέ αξίε που μας ε, παρακολουθούν και στους δύσκολες εποχές και στις καλές εποχές και σε περιόδους ειρήνης και ευημερία ή αστάθειας και προβλημάτων. Είμαστε χώρες δημοκρατικές με λαούς δημοκρατικούς, με αιρετούς εκπροσώπους και με κοινέ αξίες. Εδώ και ένα χρόνο που είμαι πρεσβευτής των ΗΠΑ δεν μπορώ παρά να πω ότι έχει ε, ενταθεί η εντύπωση που ε, είχα και πριν να έρθω για τις κοινέ αξίες που μοιραζόμαστε. Επίσης, πολλές φορές ακούγεται ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, περισσότερο ενδιαφέρονται για την ασφάλεια παρά για την προσοχή του ιδιωτικού βίου που ενδιαφέρει πιο πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σωστή αυτή η παρατήρηση. Δεν ευσταθεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε από, από τα θεμέλια τους ήδη έχουν την αρχή του σεβασμού του προσωπικού βίου. Γιατί η χώρα μας θεσπίστηκε ως μία ε, σειρά από απικίες που ιδρύθηκαν από ανθρώπους που έφυγαν από τις πατρίδες τους για να βρουν ένα χώρο ελευθερίας, προστασίας, ανεξιθρησκείας, ε, ιδιωτικού βίου. Και εδώ και δύο αιώνες έχουμε επεκτείνει και διευρύνει αυτές τις αξίες και τις ελευθερίες μαζί με τις πολύ σημαντικέ εξελίξεις και στην σύγχρονη τεχνολογία. Άρα, θεωρώ ότι είναι κοινέ και οι αξίες του ιδιωτικού βίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όμως γνωρίζουμε και εσείς όπως και εμείς ότι ασφάλεια ότι χωρίς ασφάλεια προστασία του ιδιωτικού βίου δεν μπορεί να υπάρχει. Ασφάλεια δηλαδή από την τρομοκρατική επίθεση, από τις παρεμβάσεις της τρέβλος του ανταγωνισμού και των ε, εμπορικών σχέσεων. Όλα αυτά που σημαίνουν προστασία των ελευθεριών. Και όπως είπε και η κυρία Λεμπάγη μόλις τώρα, έχουμε κοινέ αξίες με διαφορετικές προσεγγίσεις πιστεύω. Σε αυτό νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι η συμφωνία ομπρέλα την οποία διαπραγματευόμαστε ουσιαστικά έχει να κάνει με διαφορετικές προσεγγίσεις για τον ίδιο στόχο. Η ειλικρινή μας τοποθέτηση είναι ότι τις προκλήσεις πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Δεν θα πρέπει να θυσιαστεί στο βωμό της ασφάλειας ο ιδιωτικός βίος και προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να εξασφαλίσουμε και τα δύο και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τα δύο και πρέπει να συζητήσουμε, όπως πει και η κυρία Νετφέλντ, ανοιχτά και τα δύο γιατί είναι δύο του ίδιου Και βεβαίως θα πρέπει αυτό να το πράξουμε σε ένα ε, διεθνές ένα κλίμα ε, που μεταλλάσσεται διαρκώς με το ίντερνετ, με την παγκοσμιοποίηση, με το διεθνοποιημένο έγκλημα, την, το υπερσυνοριακό έγκλημα, την παιδική πορνογραφία και τα άλλα αντίστοιχα προβλήματα. Βέβαια, Καλό είναι ότι υπάρχει κοινή ιστορία και επιτυχή συνεργασία. Είχαμε καλή ε, αστυνομική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό μεταξύ μας, ΗΠΑ και Ένωση, με πολύ θετικά σημεία και επιτυχίες με προόδους σημαντικές ως προς την ε, εφαρμογή, επιβολή δηλαδή του νόμου, αλλά και ταυτόχρονα προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και για ένα παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω ότι εφέτος υπό τον τίτλο της ε, αμοιβαίας συνδρομή και απέλαση με τις 54 ε, συμπληρωματικές συνοδευτικέ συμφωνίες τους η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ συνήψαν μια συμφωνία που δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε από κοινού το οργανωμένο έγκλημα. Κοινέ λοιπόν προσπάθειε και με τη Eurojust και με τη Europol συνεργασία που επιτρέπει να ε, διερευνηθούν περιπτώσει παιδική προγραφίας ε, και παιδεραστία που μας επέτρεψε μάλιστα από την περίπτωση ενός μόνο παιδεραστή που συνελήφθη σε ένα κράτος μέλες, μέλος να μπορέσουμε να αποδιαρθρώσουμε ένα μεγάλο δίκτυο σε 25 και χώρες με τελικό αποτέλεσμα ότι σώσαμε από τα νύχια αυτού του, δι... του κυκλώματος 50 παιδιά. Πολλές άλλες είναι οι ε, περιπτώσεις συνεργασίας, η, ε, περίπτωση, η περιπτώση παραδείγματι συλλήψεως ε, φυγοπίνων και άλλων ε, διώξεων εγκλημάτων. Έχουμε συνεργαστεί σε επίπεδο ε, των καλύτερων εμπειρογνωμόνων μας μέσα από μια πολύπλευρη ε, προσέγγιση με αρχές ανακριτικές και διοκτικές, ειδικού του διεθνούς δικαίου, ανθρώπους που ε, κατέχουν κάθε είδους έννοια και ε, διαφορετικά συστήματα στο ε, δίκαιο της προστασίας των ανθρωπινών δικαιωμάτων του ιδιωτικού βίου κυρίως και με την καθοδήγηση των Υπουργών Δικαιοσύνης μπορέσαμε χάρη στην εργασία αυτής της ομάδας να καταλήξουμε σε μια δεσμευτική νομικά συμφωνία ως προς το πλαίσιο της προστασίας του ιδιωτικού βίου. Χαίρομαι λοιπόν εκ μέρους των ΗΠΑ, διότι βλέπω ότι συνεχίζεται αυτή η δουλειά, δεν έχουμε ε, να κάνουμε με το πέρας μιας διαδικασίας, αλλά με την εκκίνηση μιας διαδικασίας συνεργασίας, και όπως είπε και ο κύριος Τεκλέρκ, είναι μια απαραίτητη ε, πορεία αυτή η διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορούμε να μεταπηδούμε από τη μία συμφωνία στην άλλη. Πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση στηριζόμενη στις κοινέ μας αρχές. Ξεκινούμε λοιπόν τη δικασία των διαπραγματεύσεων και έτσι θα ήθελα και εγώ να διατυπώσω κάποιε από τι ανησυχίε που τρέφουμε από πλευρά των ΗΠΑ Η προτινόμενη εντολή λοιπόν μας γεννά ανησυχίε προ τα εξή. Θέλουμε καταρχά να είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για θέσει οι οποίε είναι σύμφωνε με τι κοινέ αρχέ πάνω στι οποίε εργαστήκαμε για να καταλήξουμε συμφωνία επί τρία χρόνια. Ένας από τους τομείς που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και προκαλεί ανησυχίε είναι η δυνατότητα της αναδρομικής ενδεχομένω δέσεως σε ισχύ αυτή τη συμφωνία. Δεν θέλουμε δηλαδή να τεθούν ένα αμφιβόλο ενδεχομένως και εκατοντάδες συμφωνιών ε, διευθετήσεων, ρυθμίσεων που έχουν περάσει από κάθε στάδιο επεξεργασίας στη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Έχουμε πολύ, επιτυχημένες, ε, πολύ επιτυχημένη συνεργασία και πολύ καλές επιδόσεις στο πεδίο αυτό μέχρι τώρα και δεν μπορούμε ε, να δεχθούμε αναδρομική ισχύ αυτής της συμφωνίας. Η συμφωνία δεν θα πρέπει να έχει τέτοια αναδρομική ισχύ που θα οδηγήσει σε περικοπή της λειτουργίας, ε, ε, ανατροπή των αποτελεσμάτων τελειπά των μέχρι τώρα συμφωνηθισών αρχών. Οι συμφωνίες που έχουμε μέχρι τώρα ούτω ή άλλως έχουν κάποια ημερομηνία λήξεω, θα ανατραπούν, θα λήξουν και μετά μπορούν να ε, ενταχθούν σε αυτή τη συμφωνία πλαίσιο, την ομπρέλα όπως λέμε. Αυτό το λέω όχι μόνο για λόγους ε, θεωρητικούς αλλά και για πρακτικούς λόγους. Φανταστείτε τι είδους επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στο δικαστικό μας σύστημα. Το να ε, επιβληθεί αναδρομική εφαρμογή ε, της νέας συμφωνίας θα οδηγήσει σοβαρά προβλήματα το δικαστικό μας σύστημα, θα ανατρέψει ακόμη και καταδίκες τις οποίες έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Οι δικαστικές αρχές από κάθε πλευρά του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ασχοληθούν και να ανοίξουν παλιούς φακέλους δίκες κατά με αβεβαιότητα φυσικά νομική που θα επικρατήσει και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να, στο οποίο δεν θα πρέπει να υποπέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θέλουμε να υποπέσουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι καλή συνεργασία, η ιστορία αυτή που έχουμε συνεργασίες μεταξύ μας, οι καλές σχέσεις θα επιτρέψουν να βρεθούν δημιουργικές λύσεις και να προχωρήσουμε. Επίσης, πιστεύουμε ότι προκειμένου να φέρει καρπούς πράγματι αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, μια δήλωση καλής συνεργασίας μεταξύ των καθεστώτων περί προστασίας του ε, προσωπικού ε, χώρου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση μια συμβατότητα μεταξύ των καθεστώτων που έχουμε για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο βαθμό του δυνατού αυτή η Γενική Συμφωνία. Έτσι λοιπόν μέσα από τη διαδικασία της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου έχουμε μπορέσει να γνωρίσουμε καλύτερα ένα τον άλλον τα καθεστώτα περί προστασίας του ιδιωτικού βίου που γνωρίζουμε, γιατί και πώς έχουμε τις ίδιες αξίες ε, και αρχές που εφαρμόζουμε ενδεχομένω κατά διαφορετικούς τρόπους δεν φρονούμε ωστόσο ότι υπάρχουν σοβαρά δυσκολίε, ούτε από την πλευρά του ενός, ούτε από την πλευρά του άλλου, δηλαδή ευρωπαϊκού ή αμερικανικού συστήματος για την προσέγγιση του προσωπικού βίου. Πιστεύουμε ωστόσο ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, να την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική και εν τέλει να προσδιορίσουμε μια κοινή αρχιτεκτονική, ένα πλαίσιο κοινό ε, για να προχωρήσουμε και να έχουμε πιο απρόσκοπτη συνεργασία. Για να, κλείνω, λοιπόν, για να κλείσω λοιπόν, θα ήθελα να τυπώσω μια πρόταση για το πώς μπορούμε εμείς, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η δική σα ιδιαίτερα ε, Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσουμε στην παρέτερο συνεργασία. Θα ήθελα να δεσμευτούμε όλοι, ιδιαίτερα τα μέλη τη Επιτροπή σα και το προσωπικό τη να συνεχίσουμε την διαδικασία εκμάθησης. Είχαμε ήδη πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ΗΠΑ. Υπήρξαν πολλά μέλη της Επιτροπής σας που μπόρεσαν να έρθουν στις ΗΠΑ να συναντηθούν με εμά, με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ή του Κογκρέσου. Είναι μια συνεργασία αυτή πιστεύω που θα πρέπει να συνεχιστεί. Και επίσης ε, και εμείς είχαμε την ευκαιρία να, ενημερωθούμε, να ενημερωθούμε από πλευρά διαφορών υπηρεσιών των ΗΠΑ αρμόδιων ε, για τα θέματα της ε, ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων και του ιδιωτικού βίου. Ο κύριο Δεκαπιτάνη μου είπε μόλι τώρα ότι ίσω η Επιτροπή σα να επισκεφθεί τι ΗΠΑ στο εγγύ μέλλον. Πράγμα στο οποίο προσβλέπουμε και εμεί με πολύ ενδιαφέρον, γιατί ασφαλώ θα εμπλουτίσει το έργο σα το να έχετε περισσότερε γνώσει για το δικό μα σύστημα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σα ζητήσω, που μπορούμε να κάνουμε μαζί δηλαδή, είναι το εξή. Μην επισκεφτείτε μόνο τι ΗΠΑ, μην αφιερώσετε δηλαδή μόνο χρόνο να μιλήσετε με τους ειδικού ε, για, την προσφυγή του ιδιωτικού βίου όταν έρχεστε εδώ, όταν έρχονται μάλλον εκείνοι εδώ οι Αμερικανοί ειδικοί, αλλά στις ε, εκλογικές σας περιφέρειες, δώστε λίγο χρόνο να μιλήσετε με τους ειδικού στη χώρα σας, ε, στην ανταλλαγή δικαστικών και αστυνομικών ε, στοιχείων, συνεργασία κτλ. Για να δείτε και εκείνοι πώ εκτιμούν τη συνεργασία με τι αντίστοιχε αρχέ των ΗΠΑ και δείτε τι σημασία έχει αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Νομίζω ότι για να καταλήξω είναι η στιγμή τώρα να αξιοποιήσουμε την κοινή μας, ε, τις κοινέ μας αρχές και αξίες. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά εν τέλει έχουμε πολλά κοινά. Πολύ περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν και θα ήθελα για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσω την κοινή μας δέσμευση στην προστασία όχι μόνο της ασφάλειας του πολίτη, αλλά και του ιδιωτικού του βίου. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να δει συγκρίνοντας τα συστήματα και νομίζω ότι αυτό το οποίο μας κάνει να ζηλεύουμε ένα τουλάχιστον από αυτά είναι το Freedom of Information Act, ο νόμος για την ελεύθερη πληροφόρηση. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει λίγο συνάδελφοι και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω από τον εισηγητή αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο και μετά θα υπάρξει μια παρέμβαση αναπολιτική ομάδα. Ήδη δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, θέλει κάποιος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το λόγο. Πείτε μου όταν τελειώσει ο ομιλητής, ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ για αυτό τον πρώτο γύρο, σας ευχαριστώ για τις ομιλίες σας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι πράγματι συμμεριζόμεθα ορισμένες ανησυχίες και επιθυμούμε να προχωρήσει και να εμβαθυνθεί η συνεργασία μας γύρω από τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του τρόπου προστασίας τους. Η ερώτησή μου είναι η εξής. σχετικά με αυτά τα οποία είπε ο κ. Κένεφ για τις υπάρχουσες μορφές συνεργασίας. Ανησυχεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο γιατί θέλει γρήγορα να αποκατασταθούν κάποια επίπεδα προστασίας των αρχών οι οποίες μας διαπνέουν, αλλά να συζητηθούν ήδη ορισμένα θέματα τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο συμφωνία στο παρελθόν στα πλαίσια της προσπάθειας συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς θα θέλαμε να υπάρξει ένα συνολικότερο πλαίσιο συζήτησης, επίπεδο συζήτησης. Και έτσι μόνο τότε θα μπορέσουμε να καλύψουμε τα κοινά, τα κενά τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να διορθώσουμε, θέλουμε να καλύψουμε. Θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε αποφασίσει να αντιδράσουμε με διαφορετικό τρόπο στις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείε και είχαμε πει ότι χρησιμοποιούνται νέοι τρόποι συνεργασίας και στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων και ταυτόχρονα Ε, εμπιστευόμεθα τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε στο μέλλον για τη βελτίωση των συστημάτων μας. Τα συστήματά μας, επαναλαμβάνω, ε, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Και πριν περάσουμε σε δεσμευτικές συμφωνίες, θα πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του αμοιβαία. Οι συζητήσεις σχεδόν έχουν κλείσει 10 χρόνια γύρω από τα θέματα αυτά και νομίζω έχει έρθει η στιγμή να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ανασχηματίσουμε προς το καλύτερο τα υπάρχοντα πλαίσια συζήτησης και προστασίας. Αυτό είναι μία από τις βασικές ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όταν συζητάμε τα θέματα αυτά με άλλες κυβερνήσεις, για την ανάγκη δηλαδή ύπαρξης ενός ευρυτέρου πλαισίου συζητήσεων. Ο κύριος Λαμπρινίδης για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ. Η ερώτησή μου απευθύνεται προς τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε συναντηθεί και σε αυτά που είπε ο Γιάννη. Κύριε πρέσβη, ανησυχώ για το εξής. Υπάρχουν εκατοντάδες συμφωνίες διμερείς ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ένωσης και της ΕΠΑ και συμφωνίες πολυμερείς ανάμεσα στην Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Η δική σας πλευρά θεωρεί ότι μια νέα συμφωνία πλαίσιο μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω σύγχυση και προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή των υπαρχουσών συμφωνιών. Από ό,τι καταλαβαίνω, στα πλαίσια των εκτιμήσεών σας, οι υπάρχουσες συμφωνίες περιλαμβάνουν κάποιους κανόνες προστασίας δεδομένων, που ίσως να διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που συζητάμε σήμερα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης συμφωνίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα ήθελα οι γραφειοκρατικές δυσκολίες που θα προκληθούν από την τροπολόγηση την οποία θα χρειαστεί να κάνουν οι ΙΠΑ να οδηγήσουν στην αποτυχία του εγχειρήματο. Εάν από την άλλη οι Ηνωμένε Πολιτείε συμφωνούν με τα θέματα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής της συνολικής, νομίζω ότι θα υπάρχει η δυνατότητα δεν θα είναι πολύ δύσκολο με την τροπολόγησή τους, ε, ίσως προσθέτοντας μία ρήτρα λέγοντας ότι οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται ανοιχτά σε σύγκρουση με τη νέα ευρύτερη συμφωνία πλαίσιο. Αν δεν το κάνουμε τότε θα υπάρξει σύγχυση, θα υπάρχει μια συμφωνία ομπρέλα για εκατοντάδες ε, επιμέρους συμφωνίες στις οποίες θα ισχύουν εντελώς διαφορετικοί κανόνες. Πώς μπορεί κανείς να έχει ένα ή οδήποτε επίπεδο ασφάλειας νομικής με την παράλληλη διάρκεια ισχύω όλων αυτών των συμφωνιών. Μπορούμε λοιπόν να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και μπορούν οι ΙΠΑ να είναι σχετικά πιο ευέλικτες γύρω από αυτό. Πρέπει να κλείσετε λέει η Πρόεδρος, θα κλείσω λέει ο κ. Λαμπρινίδης, έχετε φτιάξει ένα κατάλογο όλων αυτών των εκατοντάδων συμφωνιών και θα μπορούσατε βοηθώντας μας να μας υποδείξετε τον κατάλογο αυτών των συμφωνιών που προϋπήρχαν πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη νέα συμφωνία πλαίσιο. Κοιτάξτε σας προτείνω εφόσον συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες Υπάρχουν τέσσερις που έχουν ζητήσει το λόγο ακόμα. Ας περιμένουμε να ακούσουμε όλες τις ομιλίες και μετά θα δώσουμε το λόγο στους προλαλήσαντες. Αλλά θα ζητήσω από τους συναδέλφους μου να είναι σύντομοι γιατί έχουμε μείνει πίσω. Μπούσουτιλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια αντίδραση περισσότερο παρά μια ερώτηση. Εγώ τουλάχιστον δεν νιώθω πολύ άνετα με τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε σε αυτή την υπόθεση όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Ξεκινήσαμε καταρχήν με μια ειδική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά μιλάμε για μια γενική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα θα αναθεωρήσουμε το δικό μας νομικό πλαίσιο, το εσωτερικό. Έχω την αίσθηση ότι κάνουμε στραβά τα πράγματα, ανάποδα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας διαβεβαιώσει ότι κάνουμε το σωστό. Όσο δεν έχουμε βάλει τάξη εδώ σε εμά πώς θα μπορέσουμε να έχουμε διαπραγματεύσει με τρίτε χώρες. Τώρα για τις ΗΠΑ και προς τον κύριο Πρέσβη. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αλλαγή προσέγγισης των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια. Πριν από ένα χρόνο είχαμε την αίσθηση ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε καλά, καλά δεν ξέραν ότι υπήρχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, τώρα το ξέρουν και χαιρόμαστε γι' αυτό. Επίσης χαίρομαι πολύ κύριε Πρέσβη για τη δικιά σας προσωπική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Ξέρω πόσο σκληρά έχετε δουλέψει γι' αυτό. Κατόπιν τούτον όμως. Νομίζω ότι η συμφωνία SWIFT που εγκρίναμε θα είναι μια δοκιμή. Όχι μόνο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και πώς θα προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις για νέα θέματα, αλλά και για το πώς θα τεθούν σε εφαρμογή οι συμφωνίες μας. Θα δούμε δηλαδή με ποιον τρόπο εφαρμόζουν τη συμφωνία SWIFT Ηνωμένε Πολιτείε και αυτό θα μας διδάξει μας πολλά για τον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε εσείς τις διαπραγματεύσεις σας για την εφαρμογή άλλων ε, συμφωνιών. Εδώ άκουσα τι είπε ο κύριος ε, Λαμπρινίδης. Όντως πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο ελαστικοί όσον αφορά αυτές τις διαπραγματεύσεις. Βλέπετε, δεν θα είναι εύκολο αν δεν είσαστε ελαστικοί να προχωρήσουμε καλά. Το ξέρετε εξάλλου. Σέμον, ναι, καλά τα λες. Αλεξάνδερ Άλβαρο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Τεκλέρκ που ήρθε εδώ, όπως επίσης και τον πρέσβη των ΗΠΑ. Χάρηκα πολύ που άκουσα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, έχω δύο ερωτήσεις προς τον πρέσβη, καταρχήν. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να βάλουμε από την, άλλη μεριά, από την μια μεριά την ασφάλεια και από την άλλη μεριά τον ιδιωτικό βίο, διότι τα δύο είναι αλληλένδετα. Το ένα εξυπηρετεί το άλλο. Δεν πρέπει να τα βάλουμε σε αντιπεράθεση. Πώς να σας το πω. Δεν είναι ότι όσο πιο πολύ έχουμε το ένα, τόσο λιγότερο έχουμε το άλλο. Η ελευθερία έτσι κι αλλιώς μπαίνει πριν από την ασφάλεια. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια πολιτική άποψη. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον πρέσβη να επαναλαμβάνει αυτά που έχει πει και ο πρόεδρός σας, που είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύουμε τους πολίτες από κάθε απειλή, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο, ώστε να συνάδουν οι αποφάσεις μας και οι πράξεις μας με τους νόμους. Τελικά, legal and legitimate είναι οι δύο όροι που χρησιμοποίησε ο πρόεδρός σας τι είναι νόμιμο, τι είναι νομοταγές. Θα ήθελα να μας πείτε ακριβώς πώς βλέπετε εσείς ε, αυτή τη ε, διαφορά. Πότε γίνεται αυτό σκοπός των νομοταγές και πόσο αποτελεσματικοί μπορούμε να είμαστε. Πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα καλά. Για πείτε μας λοιπόν πού είναι το όριο ανάμεσα στα δύο. Και το δεύτερο ερώτημά μου, το είπε λίγο πολύ και ο Σέμον Μπούσιτ. Εμείς αναθεωρούμε τη δικιά μας ατζέντα όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στα μέσα της επόμενης χρονιάς φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει κάτι. Και ο συνάδελφος Άλβορθ επίσης δουλεύει για τη συμφωνία αυτή για την προστασία των δεδομένων. Και στι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης προετοιμάζεστε για μια ομοσποδιακή συμφωνία. Τελικά η συμφωνία αυτή τι θα είναι, θα είναι ένα safe harbor, θα είναι δηλαδή ένα καταφύγιο κατά κάποιο τρόπο. Θα υπάρχει κάτι ειδικό για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης ή όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταβάρες και μετά ο κύριος Γκρότσερ. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με κάτι που είπε ο κύριο Πρέσβης. Φυσικά και έχουμε διαφορετικά νομικά πλαίσια. Εδώ είμαι. Και συμφωνώ ότι τα διαφορετικά νομικά πλαίσια τηρούν τις ίδιες αρχές. Αλλά όσον αφορά τις διαδικασίες, τους στόχους ή τις δικαιωτικές διαδικασίες, τα πράγματα μπορεί να διαφέρουν. Και αυτό έχει σημασία. Όπως είπατε, πρέπει να αναγνωρίζουμε αμοιβαία τα συστήματά μας και να μελετάμε τις διαφορές. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες των Ηνωμένων ε, Πολιτειών ότι η συμφωνία, η Γενική Συμφωνία ε, δεν ε, αρκεί, γιατί υπάρχουν και άλλες τομικές συμφωνίες προηγουμένως. Εμείς θέλουμε αυτή τη Γενική Συμφωνία ε, να τις δώσουμε την ίδια τουλάχιστον ε, σημασία ιεραρχικά σαν τις προηγούμενες. Ορισμένες από έχουν επικυρωθεί και από τη Γερουσία. Θα έπρεπε και αυτή η συμφωνία να συμφωνηθεί στη Γερουσία. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ένα από τα πιο βασικά ζητήματα εδώ είναι η αναγνώριση, η μη αναγνώριση δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ανεξαρτήτως προέλευσης. Αυτό νομίζω θα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λύσουμε μεταξύ μας για να συμφωνήσουμε πάνω στο ίδιο πράγμα. Τι λύση θα μπορούσαμε να βρούμε γι' αυτό. Σίγουρα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ίσως χρειάζεται διακοινοβουλευτικός διάλογος για να δούμε τελικά τι λέει η νομοθεσία στις δύο πλευρές και τι τροποποίησεις πρέπει να επιφέρουμε στην νομοθεσία αυτή. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής, ο κ. Μπρόνς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προβλέπετε συμφωνία να ισχύει στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ή μόνο θα τηρείται από τα δικαστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ηθικά θα ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όσον αφορά τις πληροφορίες για άτομα που είναι ύποπτα για εγκλήματα που είναι εγκλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει η ελευθερία του λόγου. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, διώκεται αυτό. Ο κύριο Ντεκλέρκ είπε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που φυλάσσονται. Υπάρχουν εξαιρέσει σε αυτό. Και τέλος, τι πληροφορίες ε, ε, θέλετε να υπάρχουν ε, όσον αφορά άτομα τα οποία ειρηνικά διαμαρτύρονται, σε αντίθεση με τα άτομα τα οποία βία διαμαρτύρονται. Εμείς ακούσαμε για την τρομοκρατία, για τις και παιδεραστή και τα λοιπά. Εγώ θα ήθελα να ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε πια να σκεφτούμε και άλλες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις εκτός από αυτές τις δύο στις οποίες αναφερθήκατε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν τόσο σύντομος. Θα παρακαλέσω τους ε, ομιλητές να απαντήσουν, αλλά με την αντίστοιχη πλέον σειρά, ο κύριος Κενάρτ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω τις απαντήσεις. Ο κύριος Όλμπριχ. Στην ερώτηση για ένα ε, συνολικό πλαίσιο. Ο στόχος νομίζω είναι να συνεχιστεί η πρόοδος που έχουμε και να, να συνεχιστεί η όθηση που έχουμε λίγο πολύ εξασφαλίσει με την ομάδα υψηλού επίπεδου. και γι' αυτό δεν θέλουμε να ε, προχωρήσουμε στην αναδρομική εφαρμογή της συμφωνίας, γιατί πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε ανατροπή των αποτελεσμάτων, εάν χρειαστεί ιδιαίτερος να ε, καταγραφεί το σύνολο των συνεπειών ε, από την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής σε όλες τις δίκες και καταδίκες που έχουμε. Και για εσάς κύριε Λαμπρινίδη το ίδιο. Θα ήθελα να πω ότι έτσι όπως έχει κατασταθεί τώρα έχουμε πρακτικά το εξή πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που έχουν αυτές οι συμφωνίες μέχρι τώρα και δεν ε, θέλω να ακολουθήσω την επιχειρηματολογία ότι αποκλίνουν, όπως είπατε εσείς, ε, από τις βασικές αρχές της κατάλληλης προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων. Εμείς δεν γνωρίζουμε αν ισχύει αυτό. Από τη δική μας προοπτική, έστω υποκειμενική, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποιο ιστορικό κατάφορων παραβιάσεων του των αρχών προστασία του ιδιωτικού βίου από τι διάφορε συμφωνίε που έχουμε θεσπίσει. Αν υπήρχε τέτοιο ιστορικό, ίσω να ήταν διαφορετική η προσέγγιση μα ως προ την αναδρομικότητα τη εφαρμογή τη νέα συμφωνία, τη εντολή μάλλον. Πάντως, θα πρέπει, νομίζω, οποιαδήποτε σχετική κρίση για τον θα πρέπει να ασχοληθούν οι δικηγόροι, να εξετάσουν με ενδεχόμενο μια ανδρομική ρήτρα κτλ. Αυτό θα πρέπει να τα αφήσουμε στου ειδικού που θα αναλάβουν αυτέ τι διαπραγματεύσει. Εκεί θα πρέπει να επαφηθεί η λήψη τη απόφαση. Κύριε Μπουσούτσιλ, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σα λόγια και ε, τα συγχαρητήρια για τι προσπάθειές μα να βελτιώσουμε σχέση με το Κοινοβούλιο. σα διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε. Για δε την εφαρμογή του SWIFT από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε, πιστεύω, ότι η υλοποίηση ε, για μας δεν είναι θέμα υλοποίησης από τις ΗΠΑ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς από κοινού εργαζόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για το TFTP και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε, να γνωρίζουμε πάντοτε ότι όλα τα κύρια ζητήματα που μας ενδιαφέρουν θα υλοποιούνται σωστά από τις δύο πλευρές. Και με βέβαιο ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τηρείται ενήμερο για όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε. Για την ε, ευελιξία στην οποία αναφερθήκατε, ναι, και καθώς είμαι και παλέμαχος του SWIFT πρέπει να σας πω ότι ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ευελιξία. Προσπαθεί ο κόσμος να εξηγήσει τι είναι αυτό που θέλει, πάνω σε τι θέλει να δουλέψει, τι προκλήσεις, τι δυσκολίες αντιμετωπίζει. Αυτό ισχύει και για την Γενική Συμφωνία. Είμαι βέβαιος ότι αν εξασφαλίσουμε και από τις δύο πλευρές ευελιξία θα τα καταφέρουμε. Για τον κύριο Άβερο. Άλβαρο. Μιλήσατε για μια διάκριση μεταξύ του νομικού και του νομότυπου ή του νόμιμου και του νομότυπου ή του σύνομου. Νομίζω ότι δεν έχετε άδικο σε αυτό. Αυτό νομίζω άλλωστε αποτελεί και μια αναφορά στην οδηγία για την προσχέση του ιδιωτικού βίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δηλαδή θα πρέπει να είναι και σκόπιμη και αναλογική η παρέμβαση στον ιδιωτικό βίο. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς λαμβάνουμε υπόψη στις διαπραγματεύσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπα, δεν έχουμε, είναι διαφορετικά τα καθεστώτα που έχουμε για την προστασία του ιδιωτικού βίου, αλλά δεν είναι και στατικά. Διαρκώς βελτιώνουμε, επικαιροποιούμε, αναθεωρούμε την νομοθεσία μας και μπορεί αυτό που συζητούμε τώρα σε ένα μήνα, ένα χρόνο ή και πιο μετά να, είναι, ε, να έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Εγώ έχοντας ε, εργαστεί για πολλά χρόνια και από την πλευρά την κανονιστική αλλά και από την επιχειρηματική ε, πλευρά στο χώρο των τεχνολογιών, γνωρίζω πολύ καλά ότι οι κυβερνήσεις διαρκώς αγκομαχούν και προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις τεχνολογίας και ιδιαίτερα τώρα στο τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Ε, αυτό πρέπει να το έχουμε και ως δεδομένο στη συζήτηση για την συμφωνία γιατί και η τεχνολογία και τα καθεστώτα αλλάζουν συνεχώς και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής των ε, καθεστώτων. Κύριε Άλβαρες. Ταβάρες. Ταβάρες. Με συγχωρείτε. Ε, κάνατε μια ερώτηση σχετικά με, τον, ε, με την νομοθεσία σχετικά με την προσοχή των, των προσωπικών δεδομένων και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κογκρέσου των ΗΠΑ. Για να είμαι ειλικρινή, δεν βλέπω να ξανανοίξει θέμα ε, νόμου για την προστασία του δυτικού βίου το Κογκρέσο. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλω δεν επιδιώκει η αλλω δεν επιδιωκει Ομπάμα αυτή τη στιγμή και προσωπικώ ίσω πρέπει να σα πω τη γνώμη μου ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Βλέπω βεβαίω τα επιχειρήματα τα σχετικά με την ε, νομοθεσία αυτή την Αμερικανική και το αν εξασφαλίζει το δικαίωμα της αποκατάστασης για έναν Ευρωπαίο πολίτη που ενδεχομένω έχει φυγεί. Είναι ένα θέμα το οποίο στο πλαίσιο της ε, TFTP εξετάζουμε. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση που όμως δεν μπορεί να είναι η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη και βίου. Έχω λίγο καιρό ως προσφυγής εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετοί τομείς ε, στους οποίους πρέπει, δεδομένη μια πραγματικότητα ε, σκληρή και δύσκολη τελευταία ανάλυση, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το Κογκρέσο να αναθεωρήσει κάποιο νόμο που έχει ε, εγκρίνει, που έχει νομοθετήσει. Ε, καλούμεθα πολλές φορές να βρούμε λύσεις διαφορετικέ και εδώ αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε για τον κύριο Μπρόνς. Αν μου επιτρέψετε όμως προηγουμένως να επισημάνω ότι και ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν προσφέρει την ίδια δυνατότητα αποκατάστασης ε, ζημίας ε, για τον Ευρωπαίο πολίτη, αν και εμείς θεωρούμε ότι de facto είναι η ίδια προστασία, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με τις διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή, την υλοποίηση λέει, δηλαδή, της νομοθεσίας. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες για αποκατάσταση ζημίας ε, πέραν αυτού του νόμου, όπως η παραδείγματι προσφέρεται από την νομοθεσία τη σχετική με την ελευθερία ενημέρωσης που ανέφερε η κυρία Νετφέλτ και άλλες λύσεις. Άρα ας μην ε, εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο σε αυτό το νομοθέτημα περί προστασίας του ειδικού βίου ως μόνη λύση για την αποκατάσταση μιας ενδεχόμενης ε, ε, ηθικής βλάβης ή ζημίας του πολίτη. Κύριε Μπραντς, αν έχω προφέρει σωστά τη δουλειά το όνομά σας. Εγώ έχω εργαστεί αρκετά χρόνια ως δικηγόρος και την ώρα που άκουγα την ερώτησή σα, μου φάνηκε σαν να είμαι πίσω στη νομική, φοιτητάκο, για να, αντιμετωπίζω προφορική εξέταση. Δεν νομίζω ότι δικαιούμαι εγώ να δώσω απάντηση ω προ τα νομικά ζητήματα ενό θέματο, μια συμφωνία δηλαδή που ακόμη δεν έχει ε, περάσει από τη δικασία τη διαπραγματεύση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μην δώσω καμιά απάντηση. Ελπίζω, ελπίζω αρκετά σύντομα να μπορέσουμε όταν έρθει η ώρα να τα συστήσουμε και δημερό. Ευχαριστώ τους ε, πάντες. Ζητώ συγγνώμη αν τυχόν παρέλειψα να απαντήσω κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Κύριε Δεκλέρκ. I didn't have many questions. Δεν ε, είχα πολλές ερωτήσεις εγώ. Μία ουσιαστικά είχα. αν θα υπάρχουν εξαιρέσει. Κύριε Μπρόνς, στο χρόνο που είχα στη διάθεσή μου το σκέφτηκα. Υπάρχουν αρχές χωρίς εξαιρέσει. Μα είμαστε στην αρχή των συζητήσεων και με αυτά που είπε τώρα στο τέλος ο κύριος Πρέσβης πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και πρέπει να δουλέψουμε για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Είμαστε ευτυχείς που υπάρχουν κάποιες αρχές, ότι ξεκινάμε δηλαδή με κάποιες καλές αρχές και φυσικά φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και εξαιρέσεις, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να δώσω άλλες απαντήσεις. Το βασικό είναι το ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα πλαίσιο και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα γίνει σύνδεση με τις επιμέρους συμφωνίες και ρυθμίσεις που υπάρχουν. Αυτή είναι η δουλειά Τη επιτροπή, τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μόνο, να βρούμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα στι γενικέ αρχέ, στο γενικό πλαίσιο τη νέα συμφωνία και να υπάρχει συγχρόνω και σύνδεση με τι ήδη υπάρχουσε συμφωνίε. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μα να δουλέψει και αυτό ακριβώ θα κάνουμε. Από το Δεκέμβριο πρέπει να κοιτάξουμε να το Δεκέμβριο μάλλον πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα για τη Σύνοδο του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ, κύριε Πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα προς τον κύριο Λαμπρινίδη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα αυτό που είπε και ο κύριος Πρέσβης, ότι δεν ξέρουμε η Γενική Συμφωνία πόσο θα επηρεάσει τις υπάρχουσες συμφωνίες. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πρώτα πρέπει αυτό να ξέρουμε. Και να μην παρεκκλίνουμε από τον κύριο στόχο των διαπραγματεύσεων αυτών που είναι να συμφωνήσουμε για κοινέ προδιαγραφές όσον αφορά τη μέλουσα συμφωνία μας. Όπως γνωρίζετε, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δημιουργήσουμε ένα κοινό πλαίσιο όπου οι πολίτες θα έχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας όπου και αν βρίσκονται στην Ευρώπη. Και θα ήταν παράδοξο να έχουμε μια γενική συμφωνία γι' αυτό και να έχουμε διαφορετικές διατάξεις συγχρόνως σε διαφορετικές χώρες. Αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε. Συμφωνώ και με τον κύριο Πρέσβη ότι εμείς δεν θέλουμε το χάος, δεν είναι αυτό που θέλουμε, όχι, αλλά ανάμεσα στο χάος και σε μια κατάσταση που δεν θα προσαρμόζουμε τις υπάρχουσες συμφωνίες, νομίζω ότι υπάρχει και μια μέση οδός. Στόχος μας πάντως είναι να δημιουργήσουμε αυτό το κοινό πλαίσιο όπου οι πολίτες θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπου και αν βρίσκονται στην Ευρώπη. Τώρα για τον κύριο Μπουσάτελ. Ότι συμπεριφερόμαστε κάπως αιρετικά, Δηλαδή λέτε ότι έχετε την αίσθηση ότι δεν κάνουμε τα πράγματα με τη σωστή σειρά, αλλά ανάποδα. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι σε έναν κόσμο ιδανικά πλασμένο θα τα είχαμε κάνει διαφορετικά. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε συμφωνίες στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο λόγος όμως που θέλουμε αυτό το πλαίσιο είναι ακριβώς ότι πρώτα απ' όλα Θέλουμε να αποφύγουμε το patchwork. Θέλουμε δηλαδή να συμφωνήσουμε σε προδιαγραφές που θα είναι οι ίδιες. Κάθε φορά δηλαδή που θα πρέπει να κάνουμε διαπραγματεύσεις για μια ειδική συμφωνία, να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο που είναι κοινό. Γι' αυτό το θέλουμε αυτό το πλαίσιο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την, ε, το εσωτερικό πλαίσιο για την εσωτερική προστασία. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Και παρόλο που είναι ένα πλαίσιο που θα αλλάξει κάποια πράγματα, προσαρμόζοντας τις προδιαγραφές μας ώστε να λάβουμε υπόψη μας τις αλλαγές στην τεχνολογία κτλ. Οι βασικές αρχές δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά. Τα θεμέλια δηλαδή θα παραμείνουν. Δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη αλλαγή ό,τι και αν αλλάξει, τα βασικά θεμέλια θα παραμείνουν στη θέση τους. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπως ξέρετε, η Πρόεδρος Ρέντινγκ δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη στενή συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θυμόσαστε ότι όταν η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο εντολής για διαπραγματεύσεις, συγχρόνως υποβλήθηκε στο Συμβούλιο και ήρθε η κυρία Ρέντινγκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξηγήσει ποιες είναι οι αρχές της συμφωνίας αυτής. Και ξαναήρθε και άλλες δύο φορές προκειμένου να συζητήσει μαζί σας. Άρα θα υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, έτσι όπως υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Για αυτή την τελευταία παρατήρηση θέλω να πω και εγώ κάτι, γιατί αναγνωρίζω ότι υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στο κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι εδώ πέρα μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Δεν είναι κάτι που πρέπει να δούμε σαν ένα διοικητικό. Είναι κάτι που πρέπει να συζητιέται με τον κόσμο. Τώρα μιλάω προσωπικά βέβαια, αλλά πιστεύω ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες. Δεν είναι μόνο θέμα ανάμεσα στα τρία θεσμικά μα όργανα. Τους αφορά άμεσα. Αυτή την παρατηρήση είχα να κάνω. Λοιπόν, τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους από το πάνελ που ήρθατε και συμμετείχατε σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και έτσι τελειώνει το πρώτο μέρο. Okay, I'm. Uh, Ένα λεπτό διάλειμμα για να φύγει το πάνελ αυτό και να έρθει το επόμενο. Okay, can I invite Παρακαλώ το επόμενο πάνελ να προετοιμάζεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί κάποιοι από τους πανελίστες μας, σε εισαγωγικά η λέξη, θα πρέπει να φύγουν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την δεύτερη συνάντηση, κοινέ αξίες, συνταγματικοί περιορισμοί και πιθανές κοινέ λύσεις και αναλογικότητα, δικαστικές αλλαγές και ανεξάρτητη εποπτεία και αποτελεσματική εποπτεία. Λοιπόν, αντίθετα από ό,τι λέγεται στο πρόγραμμα, θα ήθελα να δώσω τον λόγο πρώτα στον κύριο ε, να πάρει το λόγο και ε, μετά ο κύριος Ρότεμπεργκ θα πρέπει να φύγει αφού δεχθεί κάποιες ερωτήσεις γιατί θα πάει σε μία συνάντηση για ε, συζήτηση του ηλεκτρονικού απορρίτου στην Ιερουσαλήμ. Uh, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιζενφέλντ, τον κύριο Άλμπρεχτ και τα μέλη της Επιτροπής σας που είσαστε εδώ σήμερα για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ επίσης που ομιλώ πρώτος. Πρέπει να πάω γρήγορα γιατί υπάρχει μία συνάντηση για το θέμα το συγκεκριμένο στο Ισραήλ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και για τη συνετοχή του τον πρέσβη κύριο Κανάρντ, γιατί έχει σημασία στα πλαίσια του διαλόγου αυτού που γίνεται και στις Ηνωμένε Πολιτείε και η κυβερνητική πλευρά να είναι δεκτική και να ακούει τις απόψεις για τις προηγούμενες συμφωνίες και ο κύριος Κανάρντ είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Λοιπόν, εμείς τι είμαστε, το ΕΠΙΚ. Είμαστε μια ανεξάρτητη οργάνωση η οποία έχει την έδρα της στο Washington DC, ασχολείται με θέματα ιδιωτικού χαρακτήρα και προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκδώσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις μεταφορές προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τα ταξίδια πάνω από τον Ατλαντικό, και έχουμε θέσει θέματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ακόμα και πριν από το τι συνέβη το Σεπτέμβριο ε, του 2001. Ξέρετε ότι είχαν υπάρξει και, στο, και πριν από τότε προβλήματα σχετικά με αιτήματα της Αμερικανικής κυβέρνησης για στοιχεία των επιβατών που πήγαιναν στις Ηνωμένε Πολιτείε των ρυθμίσεων των λεγόμενων ασφαλής λιμένες, εις safe harbor, πάλι στα μέσα της δεκαετίας του 90 και θέματα που αφορούσαν ε, τα συστήματα μεταφοράς χρημάτων SWIFT. Υπάρχει κάποιο παράδοξο εδώ. Απαιτείται από τη μία ισχυρή προστασία προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών. Δεν είναι ένα εμπόδιο ε, το θέμα αυτό. Όταν υπάρχει ισχυρή προστασία προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να μετακινηθούν ανάμεσα στις ε, υπηρεσίες της κρατικές και ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες με την διαβεβαίωση ότι θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά για τον σωστό λόγο ε, το αντίθετο βέβαια είναι επίσης αληθές. Η απουσία ενός τέτοιου πλαισίου, οι ροές των διατραντικών δεδομένων δημιουργούν ανησυχίες γιατί οι πληροφορίες που συλλέγονται, οι προσωπικές, μπορεί να χρησιμοποιούνται για ακατάλληλους στόχους και δημιουργούνται νέες δυνατότητες για ποινικά κολάσιμες και εγκληματικές ενέργειες. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια αυτά η προσπάθεια την οποία κάνετε σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει μεγάλη σημασία γιατί τα δεδομένα που αφορούν την επιβολή της τάξης και του νόμου είναι ιδιαίτερο ευαίσθητα. Υπάρχουν θέματα που αποδόνται ποινικών, ποινικών κολάσιμα σύμπεριφορών, απειλών στην εθνική ασφάλεια και τέτοιες πληροφορίες είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να την χάνουν της υψίστης δυνατής προστασίας. Υπάρχει και ένα δεύτερο παράδοξο όμως το οποίο θα ήθελα να σας δείσω να σκεφτείτε. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων απαιτεί διαφάνεια. Εμείς όταν συζητάμε για, την, για τον ιδιωτικό χαρακτήρα δεν μιλάμε για την μυστικότητα και την εμπιστευτικότητα των στοιχείων αλλά μιλάμε και για την εποπτεία και το υπόλογο αυτών που ασχολούνται με τα στοιχεία, έτσι ώστε οι αρμόδιες δημοκρατικές υπηρεσίες να μπορούν να εφαρμόζουν τα επίπεδα της προστασίας που απαιτείται, που προβλέπονται από τον νόμο και τα στοιχεία να χρησιμοποιούνται μόνο για τον στόχο για τον οποίο συλλέγονται. Μου ζητήθηκε να αναφερθώ επίσης ε, στο θέμα των κοινών αξιών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλές ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στη ΣΥΠΑ γιορτάζουμε έτσι και αλλιώ ε, τα 30 χρόνια των ε, κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΣΑ για τα ιδιωτικά στοιχεία, τα προσωπικά στοιχεία και συμμετέχουν στον εορτασμό φυσικά και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι και γενικότερα από τη Βόρεια Αμερική. Δεν υπάρχουν διαφωνίες για τις βασικές αρχές προστασίας των δεδομένων ανάμεσα στις ε, διάφορες κυβερνήσεις μας. Πιο πρόσφατα οι ΙΠΑ χρησιμοποίησαν και το Συμβούλιο της Ευρώπης για να υπάρξει στήριξη και για τη σύμβαση του εγκλήματος των κυβερνοχώρων και το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένα άλλο πιθανό μέσο πλαίσιο που μπορεί να παρέχει επίπεδα νομικής προστασίας στις διεθνείς επαφές. Υπάρχουν ορισμένοι κρίσιμοι τομείς όμως, τους οποίους η Αμερικανική νομοθεσία πρέπει να ανανεωθεί. Και σέβομαι αυτά που είπε ο, επίτρο, ο πρέσβης κ. Κανάρντα, αλλά από την άλλη δεν δέχονται αυτά που είπε ότι οι νομικές ρυθμίσεις στη ΣΥΠΑ είναι ικανοποιητικές στο παρόν χρονικό διάστημα. Σύντομα, πού υπάρχουν προβλήματα. Πρώτον, όπως γνωρίζετε, το Privacy Act του 1994 που αφορά τη συλλογή προσωπικών υπηρεσιών από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της κυβέρνησης, σαφώς και δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με πολίτες ε, εκτός, Ευρωπαϊκ... εκτός Ηνωμένων Πολιτειών ή παράνομα Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πολλοί κανόνες οι οποίοι δεν κάνουν διακρίσεις ανάμεσα στα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα συλλέγονται. Έχουμε όμως να κάνουμε με ένα γεγονός ότι το 1974 το Κογκρέσο έκανε αυτή τη διάκριση και αντίστοιχες διακρίσεις γίνονται και στα πλαίσια των νομοθετικών ρυθμίσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο πρόσφατα όπου υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους Αμερικανούς πολίτες και τους μη Αμερικανούς πολίτες. Δεν υπάρχει όμως λόγος να ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον πρέσβη Κανάρντ ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία απλή λύση ζητώντας από το Κογκρέσο να τροπολογήσει όλους αυτούς τους κανονισμούς και αυτό θα είναι δύσκολο. Αλλά δεν είναι χαραγμένη σε λίθο η ε, ρυθμίση αυτή και μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη μας από από το Patriot Act και μετά έχουμε αλλάξει πολλές ρυθμίσεις για τα, για στοιχεία και, την τα προσωπικά στοιχεία και την προστασία των προσωπικών στοιχείων των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε τα επίπεδα στα οποία οι δημόσιες υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφαλείας και κατασκοπίας μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά ε, <clears throat> δεδομένα των πολιτών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τις οποίες έχει προχωρήσει το Αμερικανικό Κογκρέσο. Οι ανεξάρτητες αρχές από την κυβέρνηση που αξιολογούν ε, τις διαδικασίες αυτές έχουν μειωθεί και οι ελεγκτές των στοιχείων αυτών έχουν από πλευρά της δικαστικής εξουσίας μεγαλύτερων περιθωρίων. Αυτό είναι και το πρόβλημα με τον λεγόμενο πατριωτικό νόμο, το Patriot Act. Αυτό είναι κάτι που έχει άμεση σχέση με τη συζήτησή σας. Και ένα τρίτο σημείο είναι οι νέες τεχνολογίες. Πολλές νέες τεχνολογίες έχουν αυτή τη στιγμή εφαρμοστεί στον τομέα της προστασίας του νόμου. Πολλές από αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, πολλές έχουν αμφίβολη χρησιμότητα. Το πολιτικό θέμα είναι ότι πολλές από αυτές τις νέες τεχνολογίες ε, δεν υπόκεινται στον έλεγχο του νόμου, τουλάχιστον στη ΣΥΠΑ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι στα πλαίσια των συζητήσεών σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων αυτών, ακριβώς γιατί έχουμε να κάνουμε με μια νέα δυναμική που περιλαμβάνει σαν, παράδειγμα τα καινούργια σκάνερ σώματος, σαρωτές σώματος που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια, που μπορεί να είναι χρήσιμα αλλά που θα πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένες εφαρμοστικές διατάξεις που ελέγχονται από τον νόμο. Λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να συνεργαστούμε τις, ε, με οργανώσεις όπως η δική μου που ασχολούνται με θέματα και έχουν στόχους σαν και αυτούς τους οποίους έχετε κι εσείς μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο προσπαθεί να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και είμαστε και λίγο εγωιστές σε σχέση με αυτά τα οποία κάνετε. Ο λόγος είναι απλός και βασίζεται στην ιστορική εμπειρία. Όταν εσείς ξεκινάτε μία πρωτοβουλία για να σεβαστείτε τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κάνετε αυτό όχι μόνο για τους δικούς σας τους πολίτες, αλλά και για τους πολίτες του υπολείπου κόσμου. Αυτή είναι τουλάχιστον η εμπειρία που είχαμε σχετικά με την υιοθέτηση της Αμερικανικής Οδηγίας στη δεκαετία του 90. Αναγκάσατε και άλλες κυβερνήσεις να προσαρμοστούν και να διορθώσουν την ανεπάρκεια των δικών τους νομικών ρυθμίσεων. Έχετε την δυνατότητα λοιπόν να θέσετε υψηλότερα επίπεδα προστασίας των πολιτών σας και των καταναλωτών και αυτό το κάνατε και πριν από το διαδίκτυο και πριν από τις νέες τεχνολογίες που συζητάμε σήμερα. Ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια η οποία ανύψωνε τελικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό τους σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό λοιπόν είναι τιμή μου που είμαι εδώ, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσπάθεια την οποία κάνετε και θα ήθελα να τη στηρίξω. Ερωτήσεις τώρα. <laughs> Κύριος Λαμπρινίδης λέει πρόεδρος το φανταζόμουν. Με χαρά σας βλέπω εδώ κύριε Ρότεμπερκ. Τι θέλω να ρωτήσω λοιπόν, εάν συμφωνείτε με τις προφανείς ανησυχίες των ΗΠΑ, της κυβέρνησης των ΗΠΑ ως προς τις δυσκολίες που μπορούσε να ε, επιφέρει η εφαρμογή σε υφιστάμενες ήδη συμφωνίες, μιας νέας συμφωνίας ε, τύπου ομπρέλας. Ιδιαίτερα ως προς ε, τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν σε επίπεδο αγωγών που έχουν ε, ασκηθεί από ε, Ευρωπαίους ε, στις ΗΠΑ και την δυνατότητα για εφαρμογή υποχρεωτική ή μη νέα συμφωνίας η κυρία Νετφέλτ, αν μου επιτρέπετε, επειδή θέλει ο εισηγητή να διατυπώσει μια ερώτηση, να ακούσετε όλε τι ερωτήσει και μετά να απαντήσετε. Κύριο Άλμπρεχτ, θα συνεχίσω κι εγώ σε αυτή την ιδέα. μια και ακούστηκε ίσως να υπάρξει αναδιατύπωση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ίσως λοιπόν πρέπει να περιμένουμε να δούμε ε, κάποια αντίδραση από πλευράς των ΗΠΑ, κογκρέσου και λοιπόν κύκλων στα όσα πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια και ήδη έχουν ε, σημειωθεί κάποιες εξέλιξεις και στις ΗΠΑ, γιατί και για εμάς είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτός ο υπερατλαντικός, ο διατλαντικός μάλλον διάλογος. Το είπε και η Σοφή νωρίτερα, πρόκειται ένα ζήτημα ε, που ενδιαφέρει τους πολίτες και θα το συζητήσουν και οι πολίτες. Δεν αφορά μόνο δηλαδή περιορισμένους κύκλους και τους διαπραγματεύτέ. Ο κύριος Στάβαρης παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω σε αυτή την υπόθεση του νόμου, της νομοθεσίας περίπτωσης του ιδιωτικού βίου, γιατί πραγματικά εκεί έχουμε το κύριο πρόβλημα και πρόσκομα. Και πραγματικά δεν είμαι ικανοποιημένη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό οι αρχέ. Μπορεί να μα λέτε ότι δεν είναι θεόπνευστη βίβλο, αλλά πάντω φαίνεται ότι έτσι το χειρίζονται το θέμα οι αρχέ μόνο μια ίσονο σημασία τροποποίηση την οποία ζητούμε, δηλαδή αναγνώριση ισότιμων δικαιωμάτων προς τους αλλοδαπούς, δικαιωμάτων που έχουν ήδη οι κάτοικοι και ε, οι θαγενείς των ΗΠΑ, οι υπήκοοι των ΗΠΑ, υπάρχουν τόσο πολλές αντιδράσει. Ίσως ε, και σε αναφορά μετά στα όσα είπε ο κύριο πρεσβευτή, ο κύριο Κενάρτ νωρίτερα, μάλλον δεν έχει αντιληφθεί το Κογκρέσο πόσο μεγάλη σημασία έχουν όλα αυτά για μα. Διότι βέβαια, ό,τι άλλη συμφωνία και να συναυθεί δεν θα έχει καμιά αξία εάν ο Ευρωπαίο πολίτη δεν έχει ισότιμα δικαιώματα μέσα στι ΗΠΑ όπω ο Αμερικανό. Παρατήρηση αν θέλετε περισσότερο, αλλά πάντω περιμένω να μου απαντήσετε εάν βλέπετε κάποια δυνατότητα συνεργασία έτσι ώστε να εξηγήσουμε τουλάχιστον πόσο μεγάλη σημασία έχει για μας αυτό το νομοθέτημα. Ευχαριστώ, λέει κυρία Νετφέλτ, και μου επιτρέπετε θα διατυπώσω και εγώ μια ερώτηση. Η... Αυτή η συμφωνία, η Περατολική Συμφωνία για την πλησία των Δεδομένων Προσωπικού Βίου, που ε, καλύπτουν την μεταφορά ε, δεδομένων μεταξύ αρχών, δημοσίων αρχών και ενδεχομένως και επιχειρήσεων ιδιωτικών προς τις αρχές, όπως το PNR ή στο SWIFT προς τις Αμερικανικές Αρχές. Βλέπουμε ότι καλούνται οι πολίτες πολύ συχνά, φερειπίνει στο ηλεκτρονικό σύστημα για την χορήγηση άδεια ταξιδίου ή για τη θεώρηση ακόμη διαβατηρίου, να διαθέσουν τα προσωπικό τους δεδομένα χωρίς κάποιον ενδιάμεσο απευθείας στις αρχές των ΗΠΑ. Δεν μεσολαβεί δηλαδή κάποια αρχή ευρωπαϊκή. μεταξύ του Ευρωπαίου πολίτη και των Αμερικανικών αρχών. Αν καταλαβαίνω σωστά λοιπόν, αλλά θα με διορθώσει ενδεχομένω, μάλλον δεν θα καλύπτονται από μια τέτοια υπερατλαντική συμφωνία τέτοιου είδου ε, ε, δεδομένα. Αλλά θα καλύπτονταν εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα επέκταση τη νομοθεσία περιπτωσία του ειδικού βίου, έτσι ώστε να καλύπτει και του Ευρωπαίου πολίτε. Κύριο ε, Ρότενμπεργκ. Ναι, εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να απαντήσω ξεκινώντα προ τον κύριο πριν ίδιο προ την αναδρομικότητα τη εφαρμογή ε, τη ε, συμφωνία. Οι ανησυχίε σε επίπεδο ΗΠΑ είναι γνήσιε, πιστεύω. Έχουν να κάνουν με την ε, σκοπιμότητα της αναθεώρησης τέτοιου είδου αποφάσεων, καταδικών κτλ. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο, παραδείγματι, έχει καταδικαστεί από μια προηγούμενη απόφαση και τώρα θα ενημερωθεί για την θέσπιση μια τέτοια συμφωνία η οποία θα επιτρέπει την ε, ακύρωση στοιχείων αποδεκτικών που είχαν κατά τρόπο παράτυπο συλλεχθεί, θα σπεύσει να ακυρώσει τη δίκη του. Αυτή είναι η ανησυχία λοιπόν των ΗΠΑ. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε την ε, διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει αναδρομική εφαρμογή όσον αφορά ε, ήδη οριστικές συμφο... ε, δικαστικές αποφάσεις, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με τη συμφωνία ε, στις πιο πρόσφατες μόνο περιπτώσεις. Νομίζω ότι έτσι δίνεται η κατάλληλη απάντηση και στις ανησυχίες των ΗΠΑ. Για τον κύριο Άλμπρεχτ, που ρωτάει για τον νόμο περί προστασίας του ιδιωτικού βίου. Πάλι δύσκολη υπόθεση. Τέτοιοι νόμοι, ξέρετε, στι ΗΠΑ ε, δεν αναθεωρούνται εύκολα, γιατί ε, το να ξεκινήσει μια διαδικασία αναθεώρηση οδυναμεί με το να ανέχουμε του ασκού του αιώλου. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού θα πάει η αναθεώρηση, τι αντιπρόταση θα διατυπωθεί. Αλλά θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια προστασία του προσωπικού βίου με συνέπεια να, ζητηθεί από τις, να προκύψει ο Ισανάκη για τι ΗΠΑ να αναθεωρήσουν αυτή την νομοθεσία. Έμεση συνέπεια, δηλαδή, αν καταλαβαίνετε το επιχείρημά μου. Και έτσι μπορεί ως ευρύτερη προσπάθεια, όχι δηλαδή ως στοχευμένη επίθεση κατά αυτής της νομοθεσίας, προσπάθεια δηλαδή αν θεώρησε αυτής της νομοθεσίας και νομίζω ότι αυτό απαντά και στον κύριο Τάβαρες, ε, αλλά έμεσα. Ε, παραδείγματι, Η Υπηρεσία για την Εσωτερική Ασφάλεια στις ΗΠΑ έχει ζητήσει την ε, εφαρμογή του νόμου ε, περί προσθέσεων των ιδιωτικών δεδομένων, αλλά Ε, η δυσκολία έγκυται ε, ως προς την ε, ανυπαρξία, έγκυται στην ανυπαρξία μηχανισμού εφαρμογής, καταστολής, για να το πω διαφορετικά. Για την κυρία Ινετφέλτ θα ήθελα να απαντήσω επίση ότι το δύσκολο εν τέλει είναι το να θεσπιστεί ένα νομικό καθεστώς όπου θα μπορεί ο πολίτης να εξασφαλίσει εφαρμογή ουσιαστική των θεμελιωδών του δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι έχουμε καλέ αρχέ, συμφωνήσαμε πάνω σε, ένα σύνολο αρχών, καλών αρχών κτλ. Δεν αρκεί αυτό. Η δική μα η προοπτική υπαγορεύει ακριβώ την ουσιαστική υλοποίηση. Ακριβώ εκείνη η δυσκολία για μα. Είναι καλέ οι αρχέ και γι' αυτό επιμένουμε ότι, δεν, ότι θα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί. Και εκεί ακριβώ έγκυται και η δυσκολία για σας πώ θα εξασφαλίσετε την ουσιαστική υλοποίηση, εφαρμογή αυτών των τόσο καλών αρχών που έχετε εισαγάγει. Και ζητώ συγγνώμη που χρειάζεται να αποχωρήσω, αλλά δυστυχώ δεν έχω άλλο χρονικό περιθώριο. Ευχαριστώ που με δεχθήκατε. Κυρία Νετφέλτ. Ευχαριστούμε πολύ και ξέρετε, εμεί γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει ταξίδι. Συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει. Η ώρα περνάει. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε επιταχύνοντας κάπως τους ρυθμούς μας. Επόμενο στον κατάλογο είναι η κυρία Κριστίλα Κόστ, που είναι νομική σύμβουλος στην πολιτική όσον αφορά την ε, προστασία δεδομένων, στην εποπτεία προστασίας δεδομένων δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω σήμερα στην ακροασή σας. Ο Πίτερ Χούστινγκς έπρεπε να έρθει, αλλά θα συμμετάσχει μαζί με τον κύριο Ρότεμπερκ τώρα σε μια μεγάλη διάσκεψη. Γι' αυτό και δεν μπορεί να είναι παρόν. Έτσι έχω εγώ το προνόμιο και την ικανοποίηση να έρθω εδώ και να συζητήσω μαζί σας. Θα προσπαθήσω να αναπτύξω τα κύρια σημεία όσον αφορά τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ποια είναι τα κύρια σημεία που έχουμε αναπτύξει με γνωμοδοτήσεις για να απαντήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό του διατραντικού διαλόγου. Πιο συγκεκριμένα, ιστορικά, ποιος είναι ο ρόλος των αρχών προστασίας δεδομένων. Και μετά θα έρθω σε διάφορα άλλα σημεία που έχουν να κάνουν με την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα, ποια σημεία πιστεύουμε εμεί ότι πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω. Από το 2008 και μετά παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και ιδιαίτερα τις εργασίες του High Level Contact Group, της ομάδας αυτής υψηλού επίπεδου και έχουμε δημοσιεύσει γνωμοδότηση που είναι και στην ιστοσελίδα μας και συμμετείχαμε και στις ε, διαβουλεύσεις που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ομάδα των 29 ε, που συμμετέχουν οι Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων από την Ευρώπη. Θα έλεγα λοιπόν γενικά μιλώντας για τα έγγραφα αυτά τα οποία είναι δημόσια και τα οποία θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και τη δικιά μας. Εγώ να πω ότι υποστηρίζουμε ξεκάθαρα την ιδέα να υπάρχει διατλαντική συμφωνία η οποία να αντιστοιχεί στι κατευθυντήριε γραμμέ στις οποίε αναφέρθηκε η Επιτροπή και υπενθύμησε η κυρία Λεμπάγη πριν από λίγο. Στόχο είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει μια νομική βεβαιότητα όσον αφορά την προστασία αυτή και ένα ψηλό επίπεδο προστασία. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που στηρίζουμε εμεί απόλυτα και γι' αυτό στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Κάτι άλλο σημαντικό έχει να κάνει με τον ίδιο τον τίτλο του σχεδίου που επεξεργαζόμαστε. Μιλάμε για την επιβολή του νόμου, μάλλον μιλούσαμε για την επιβολή του νόμου, τώρα μιλάμε για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Άρα περνάμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο και πιο ξεκάθαρο και είναι σημαντικό γιατί όταν μιλούσαμε για την επιβολή του νόμου δεν είχαμε τα ίδια κριτήρια στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Όταν μιλάμε για μετανάστευση στις Νομένες δεν είναι επιβολή του νόμου όπως ε, το εννοούμε στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι καλό που είμαστε πιο συγκεκριμένοι τώρα. Πολύ σύντομα θα υπογραμμίσω τώρα πόσο μεγάλη σημασία έχουν για μας οι αρχές της συμφωνίας που έχουν να κάνουν με την νομιμότητα, με την αναλογικότητα, με τη διαφάνεια και με την τήρηση της αρχής που έχει να κάνει με το στόχο, με το τέλος. Όσον αφορά την αναλογικότητα, θέλω εδώ να προσθέσω ότι έχει σημαντικές συνέπειες όσον αφορά το είδος μεταβίβασης. Για παράδειγμα, συμφωνίες τύπου PNR ή άλλες που σημαίνει μαζική μεταφορά δεδομένων. Λοιπόν, το κριτήριο αυτό της αναλογικότητας είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επανέρχομαι τώρα σε τέσσερα σημεία που κατά τη γνώμη μου πρέπει να προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως. Είναι τα δικαιώματα των ατόμων, η εποπτεία, η μετέπειτα μεταβίβαση και τέλος το πεδίο εφαρμογής. Στην αρχή συζητήσαμε σήμερα για αυτά, αλλά εγώ έχω και άλλα πράγματα να υπογραμμίσω από την οπτική γωνία του Ευρωπαίου επόπτη. Η δυνατότητα προσφυγής που πρέπει να έχουν οι πολίτες όχι μόνο διοικητική όμως, αλλά και στα δικαστήρια. Δηλαδή, είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είτε πρόκειται για το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι πολίτες να μπορούν να προσφύγουν εκεί. Είναι πολύ βασικό αυτό η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Να υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένος τρόπος. Ήδη ο διάλογος με τις ΗΠΑ είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Κάτι άλλο σημαντικό για τα δικαιώματα των ατόμων είναι η δυνατότητά τους να προσφεύγουν άμεσα ή έμεσα στα προσωπικά τους ε, δεδομένα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό στα σημερινά πλαίσια, όπου λαμβάνονται αποφάσεις από την αστυνομία μερικές φορές που έχουν σοβαρές συνέπειες για το άτομο. Για παράδειγμα, ε, μπορεί να περιοριστεί η ελευθερία του, η στέρηση της ελευθερίας. Προβλέπονται εξαιρέσεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει εγγύηση αυτή που είναι έστω και η έμεση πρόσβαση των ατόμων στα προσωπικά τους δεδομένα. Τώρα στη συνέχεια, η εποπτεία από μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Το πλεονέκτημα να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή είναι ότι έτσι έχετε μια πιο άμεση αρρωγή. Αν χρειαζόσαστε βοήθεια δηλαδή την έχετε άμεσα. Άρα, από τη μια υπάρχει το θέμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη, από την άλλη υπάρχει ανεξάρτητη αρχή. Το τρίτο τώρα που μας απασχολεί είναι η παρετέρω μεταβίβαση δεδομένων. Είτε πρόκειται για την τρίτη χώρα, στην περίπτωσή μας οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε πρόκειται από αυτή τη χώρα σε μια άλλη τρίτη χώρα, πρέπει να υπάρχουν ε, δύο κριτήρια, χωρίς εξαίρεση. Το ένα είναι η αρχή του τέλους, του στόχου για τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και το δεύτερο είναι να υπάρχει εγγύηση για κατάλληλη προστασία στην άλλη τρίτη χώρα. Δεν θέλουμε καμία εξαίρεση σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Και έρχομαι και στο τελευταίο που είναι το πεδίο εφαρμογή. Και αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Εδώ, πάντα στα πλαίσια των αστυνομικών αρχών, το πεδίο εφαρμογή είναι ζωτική σημασία. Μερικές φορές διάφορες βάσεις δεδομένων δεν είναι απόλυτα στεγανές, είτε σε επίπεδο Ευρώπης είτε σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρουμε ότι μεταφέρονται τα δεδομένα πολλές φορές από μία υπηρεσία στην άλλη. Το γιατί και αυτό είναι κάτι περίπλοκο. Και έρχομαι εδώ στο θέμα της εθνικής ασφάλειας. Συζητάμε το πεδίο εφαρμογή τη συμφωνία αυτή και θέλουμε να ξέρουμε κατά πόσο εφαρμόζεται και στι περιπτώσει εθνική ασφάλεια. Αν η καταπολέμηση τη εγκληματικότητα και τη τρομοκρατία επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς πώς κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα δύο και πώς θα εμποδίσουμε να μεταφέρονται στοιχεία από μια βάση δεδομένων που έχει να κάνει με την ε, ε, ασφάλεια από την εγκληματικότητα στην ε, άλλη ασφάλεια από την τρομοκρατία. Μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία που να καλύπτει το σύνολο και με τι προϋποθέσεις. Είτε πρόκειται για την Ευρώπη, είτε πρόκειται για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πάντα είμαι στο ίδιο σημείο το πεδίο εφαρμογή. Υπογραμμίζω κάτι που για μας, για τον Ευρωπαίο Επόπτη, είναι πολύ σημαντικό. Είναι οι προηγούμενες συμφωνίες και επόμενες. Πρέπει να υπάρχει νομική ασφάλεια και τα ενδιαφερόμενα άτομα ε, να μπορούν να προβλέψουν τι θα συμβεί. Δηλαδή, πρέπει σε αυτές τις συμφωνίες να λαμβάνουν υπόψη μας και τις διμερείς συμφωνίες που καλύπτουν τους ίδιους στόχους. Τελευταίο για αυτό το θέμα, για το πεδίο εφαρμογή είναι το εξή. Το ακούσαμε ήδη εδώ σήμερα από τον κύριο Ντεκλέρκ, τον Βέλγο Υπουργό Δικαιοσύνη, το ότι πρέπει να υπάρχει ένα επιπλέον πλαίσιο με μια γενική συμφωνία που να δουλεύει σαν ομπρέλα και ειδικέ συμφωνίε κατά περίπτωση. Πράγματι, και εμείς πιστεύουμε ότι οι δικέ αυτές συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές για να υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας κάθε φορά που μιλάμε για μεταβίβαση δεδομένων. Το συζητάμε πολύ όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρει δεδομένα στο δημόσιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γενικά νομιμοποιούνται οι μεταβιβάσεις δεδομένων από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο τομέα. Είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε πολύ καλά πριν καθορίσουμε τις επιμέρους συμφωνίες. Έπειτα, οι δικές συμφωνίες δεν θα πρέπει να επιτρέπουν εξαιρέσεις στο γενικό πλαίσιο. Πάλι για να υπάρχει μια νομική βεβαιότητα και να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τέλος, επανέρχομαι και σε μια άλλη παρατήρηση που έκανε κάποιος ευρωβουλευτής. Πρόκειται για τις προθεσμίες και το timing. Και ο Ευρωπαίος Επόπτης το επισήμανε αυτό σε μια γνωμοδότησή του την προηγούμενη εβδομάδα για τα δεδομένα των επιβατών αεροπορικών εταιριών, το PNR. Πρώτα πρέπει να συζητήσουμε τις μεταβιβάσεις προς τρίτες χώρες δεδομένων και PNR και μετά να μιλήσουμε για μια γενική συμφωνία και να δούμε ένα άλλο επίπεδο στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει να υπάρχει μια συνοχή δηλαδή και μην ξεχνάμε ότι όταν συζητάμε αυτές τις διάφορες πτυχές, στόχος μας είναι τα διάφορα μέτρα να είναι συνεκτικά μεταξύ τους, είτε πρόκειται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε διεθνές επίπεδο. Uh, ε, επομένη, είναι η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Ναμύρ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι χαρά το να μπορώ να ανταλλάξω ορισμένε απόψεις μαζί σας, λέει η κυρία Γκερέλα. Πολλά θέματα καλύφθηκαν από τους προηγούμενους ομίλητες και θα ήθελα στα πλαίσια της παρουσίασής μου να επανέλθω ίσως σε κάποια θέματα που χρήζουν υπογράμμισης. Υπάρχουν αρκετές ασυμβατότητες στο ευρωπαϊκό και το αμερικανικό σύστημα και έχουν ήδη εντοπιστεί κυρίως από ακαδημαϊκούς τις μελέτες τους. Ανάμεσα στις βασικές ανησυχίες οι οποίες τίθενται από τους εμπειρογνώμονες αυτούς είναι κάποιες αρχές σχετικά με την διατήρηση των στοιχείων αυτών και την έννοια της ε, αναλογικότητας την ερμηνεία που δίδεται στη συγκεκριμένη ένωτα. Σχετικά με τον ορισμό του στόχου χρήσης. Ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει η έννοια του routine use, δηλαδή συνήθις ε, χρήση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην ευρωπαϊκή πλευρά και απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση γιατί απαιτούνται συγκεκριμένοι στόχοι οι οποίοι πρέπει να είναι συμβατοί. Αυτό είναι σαφέστατα ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος στα πλαίσια της προτινόμενης συμφωνίας. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι και από ευρωπαϊκής πλευράς η αρχή του περιορισμού των στόχου είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω γιατί οδηγεί σε μία όλο και πιο μεγαλύτερη πρόσβαση των αρχών καταστολής ε, στις, στα προσωπικά δεδομένα και αυτό δείχνει ότι δεν γίνεται απόλυτα σεβαστή η αρχή αυτή από ευρωπαϊκής πλευράς. Έχουμε λοιπόν και εμείς κάποιες δικές μας αντιφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε το απαιτούμενο επίπεδο συμφωνίας και με τους Αμερικανούς. Αυτή ήταν μια προκαταρκική παρέμβαση. Τώρα θα ήθελα να έλθω στους πραγματικούς ε, μηχανισμούς επιβολής ε, των συστημάτων προστασίας στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές μελλοντικέ συμφωνίες. Αυτό είναι το βασικό μου θέμα. Το πρώτο θέμα, και εδώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ η λέξη καταλληλότητα την οποία άκουσα σήμερα, δεν υπήρχε η λέξη αυτή ε, στην συμφωνία την αρχική, ενώ τώρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο καθίσταται πλέον σαφής στόχος. Θα ήθελα να πω ότι αν οι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, δεσμεύεται από αυτές τις, από αυτές τις ρυθμίσεις καταλληλότητας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε η ε, καταλληλότητα αυτή σε επίπεδο μεθόδου πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επίπεδο αρχής και σε επίπεδο στόχου σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση. Η καταλληλότητα σαν μέθοδος είναι κάτι το χρήσιμο και υπάρχει ένα ενδιαφέρον έγγραφο εργασίας, το υπαριθμ 12, το οποίο έχει σωρεύσει αρκετές εμπειρίες στα πλαίσια των θεμάτων του πρώτου πυλώνα. Και νομίζω ότι παρέχει ήδη μια σαφέστατη καλή βάση συζήτησης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί και στον τομέα της συνεργασίας, των αναγκών στις, στον τομέα της συνεργασίας σε θέματα ποινικά. Αλλά σχετικά με τους μηχανισμούς επιβολής έτσι όπως ορίζονται σε αυτό το έγγραφο εργασίας δεν υπάρχουν αντιφάσεις με τις ε, συμφωνίες ε, πλαίσιο με τη ΣΥΠΑ. Έχουν σαν στόχο οι ρυθμίσεις αυτές να ε, φέρουν εις πέρας τρεις στόχους. Πρώτος, υψηλό επίπεδο συμβατότητας με τις ήδη υπάρχουσες νομικές ρυθμίσεις. Στόχος βασικός πάλι της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία ανεξάρτητων αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στη ΣΥΠΑ και στην Ένωση στον τομέα αυτό. Οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες λειτουργούν σαν συμβουλευτικά σώματα και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν διαρθρωτικά ανεξάρτητες απέναντι στις Αμερικανικές αρχές. Όμως ε, ε, μια ευρύτερη προσπάθεια ανεξαρτησίας πέραν της ε, δικαστικής πρόσβασης είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να γίνει αποδεκτό σε πολλά νομικά συστήματα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είναι μείζον εμπόδιο στα πλαίσια της προσπάθειας για περαιτέρω διαρθρωτική ανεξαρτησία γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντισταθμιστεί και με άλλες εγγυήσει σχετικά με την, με την ανεξαρτησία, η οικονομική πόρη της αρχής, το κανονισμός ε, προσωπικού. Γενικά υπάρχει μια ολόκληρη σειρά θεμάτων, τομέων μάλλον, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπάρξουν εγγυήσει για το μέγιστο επίπεδο ανεξαρτησίας, αν και στο αμερικανικό συνταγματικό σύστημα είναι δύσκολο να διακόψει κανείς τον σύνδεσμο ανάμεσα στον υπεύθυνο ελεγκτή και στην συγκεκριμένη αρχή που είναι υπεύθυνη για τα θέματα προστασίας. Δεύτερος βασικός στόχος είναι η υποστήριξη και η βοήθεια που θα πρέπει να δίδεται στους πολίτες στα πλαίσια της πράσπισης των δικαιωμάτων τους. Η ομάδα εργασίας λέγει ότι θα πρέπει να μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί τα δικαιώματά του γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς υπερβολικό κόστος. Το μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής και σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων πρόσβασης του πολίτη και σχετικά με τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιεί. Όταν τα λέω αυτά είμαι ίσως εκτός θέματος, αλλά η αποτελεσματικότητα της άσκησης της προσωπικής προστασίας ε, ε, σαν παράδειγμα ενός πολίτη στις Ηνωμένε Πολιτείες όταν δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει τα κατάλληλα έντυπα, όταν δεν ομιλεί την αγγλική κτλ. Είναι ουσιαστικά πρακτικά εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων του καθενός. Θεωρώ λοιπόν ότι οι αρμόδιες αρχές εδώ θα πρέπει να εμπλέκονται θα πρέπει να παίζουν τον ρόλο του interface ε, ανάμεσα στον πολίτη, στον επιβάτη πολίτη και στην κυβέρνηση, στις κυβερνητικές υπηρεσίες. Αυτό θα επιτρέψει τη δυνατότητα έβρεσης έμεσων τρόπων προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να αντιμετωπίσω σαν παράδειγμα την αίτηση πρόσβασης, το access το λεγόμενο. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να το συμπληρώσει κανείς. Δεν ξέρω αν εσείς το κάνετε με πιο επιτυχημένο τρόπο από μένα, αλλά είναι δύσκολο. Εμένα μου απάντησαν ότι η αίτησή μου ε, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, αλλά ούτε και να απορρευθεί, να απορριφθεί, συγγνώμη, γιατί δεν είναι σαφές αν ε, έχει αναγνωριστεί η υποψηφιότητά μου από το FBI. Νομίζω λοιπόν ότι ε, στην ουσία μιλάμε για την κορύφωση της συνεργασίας της αστυνομικής και της δικαστικής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι δύο πλευρές την ίδια κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί. Αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι το θέμα της αποζημίωσης, αν υπάρχουν προβλήματα, αλλά και της δυνατότητας δικαστικής επανεξέτασης και αποκατάστασης παραβιάσεων ε, των ε, αρχών, από πλευράς των αρχών των προσωπικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι δόθηκαν αρκετές εξηγήσει οι οποίες δείχνουν ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί εποπτεία η οποία προηγείται τη συλλογή των στοιχείων στα πλαίσια των ποινικών διαδικασιών, στην ουσία εξαιρεί ορισμένα στοιχεία. Και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα όχι μόνο της αποκατάστασης, αλλά γενικότερα της δικαστικής επανεξέτασης όλων αυτών των θεμάτων. Λυπάμαι που σας έκοψα το λόγο, αλλά έχουμε πολύ περισσότερους ομιλητές. Τώρα ο κύριος Πάτρικ Μπράιερ, παρακαλώ, από την Ομάδα Εργασίας για την ε, Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων, σχετική δηλαδή υπηρεσία της ε, ε, Γερμανίας και εκφράζει με την ομιλία του ένα δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων δραστήριων στο τομέα αυτών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για, τη, για τα ευγενικά σας λόγια. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Ιδιαίτερα εκτιμώ το γεγονός ότι υπογραμμίζετε την ανάγκη να γίνει ο διάλογος δημόσια στην υπόθεση αυτή και ελπίζω να μπορέσω και εγώ να συμβάλλω. Εδώ αν δείτε την ε, φωτογραφία που έχω περιλάβει στην πρώτη μου διαφάνεια, πρόκειται για μία ε, πορεία διαμαρτυρίας ε, στην, ε, που έλαβε χώρα εφέτος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την παρακολούθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν το προσωπικό βίο με τρίτε χώρε όπω οι ΗΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν ξεκινώντα να αναφερθώ στα δεδομένα και τι επιδόσει των ΗΠΑ ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα για να ανοίξουμε τη συζήτηση στο θέμα αυτό. Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ στι υποχρεώσει ε, τι σχετικέ με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη δυνάμει των ισχυουσών συνθήκων και τρίτον τα τρία στοιχεία που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί ισοδύναμο επίπεδο προστασίας από τις δύο του Ατλαντικού. Ξεκινώντας λοιπόν με τις επιδόσεις των ΗΠΑ ως προς, τις, ε, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει συστηματική παραβίαση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεχιζόμενη. Δεν χρειάζεται να επισέλθω στις λεπτομέρειες. Είναι γνωστά τα δεδομένα, αναγνωρισμένα και από διεθνείς ε, φορείς όπως η ε, Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως ο ειδικό Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο κ. Σάρενινγκ. Ε, το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι όλα αυτά τα προβλήματα σε σχέση με την ανταλλαγή των πληροφοριών. Δηλαδή, όταν γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών με μια τρίτη χώρα που τακτικά και συστηματικά παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαθέτοντάς της τα στοιχεία αυτά, εξασφαλίζεται την πιθανότητα ή τη δυνατότητα να καταχραστεί τις πληροφορίες αυτές η τρίτη χώρα για παραβίαση των δικαιωμάτων. Όταν υπάρχει δηλαδή συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεννάται με τον τρόπο αυτό ο κίνδυνος για ενίσχυση αυτών των παραβιάσεων. Παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή Αρχή Καταπολέμησης των ε, Εγκλημάτων της Γερμανίας διέθεσε στοιχεία για τον Γερμανό πολίτη, τον κύριο Ζαμάζ, για το που βρίσκεται, που κατοικεί, διαμονή κτλ. με τι ΗΠΑ. Οι οποίοι στη συνέχεια τον συνέλαβαν σε άλλη χώρα, τον παρέλαβαν ε, πράκτορες της CIA, τον μετέφεραν στην Συρία, όπου υπέστη βασανιστήρια και ε, κράτηση χωρί απαγγελία κατηγοριών. Όταν απελευθερώθηκε, ε, όταν αποφυλακίστηκε, προσπάθησε να προσφύγει στα ε, αμερικανικά δικαστήρια για να ε, ασκήσει αγωγή κατά των ΗΠΑ, όπου όμως δεν μπόρεσε να δικαιωθεί διότι ε, υπερίσχυσε η νομοθεσία σχετική με το απόρριτο των πληροφοριών που διτείνεται από τις σχετικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την προστασία του ιδιωτικού βίου μόνο, αλλά με την προστασία της ελευθερίας ή προστασία από φυλάκιση παράνομη κράτηση, αλλά πολλές φορές ε, τίθεται και ζήτημα ζωής ή θανάτου. Γι' αυτό μιλούμε με τόση έμφαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι, πληροφε... οι υποχρεώσεις λοιπόν, τις οποίες έχει αναλάβει η Ευρώπη και που έχει όταν προσφέρει τις πληροφορίες, είναι σαφής η καθοδήγηση των δικαστηρίων. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κράτος το οποίο σημαίνει πραγματικό κίνδυνο παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν μπορεί κανείς να συμπράττει ε, σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από, κάποιο τρίτο κράτος. Αντιθέτω, εάν πρόκειται για ένα κράτο το οποίο διαφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και, και προσφέρει ουσιώδεις εγγύησει και μηχανισμούς ελέγχου της στήρησης αυτών κατά τρόπο ισοδύναμο με αυτόν που προβλέπει η σύμβαση, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα δηλαδή, τότε είναι δυνατή συνεργασία. Αυτά είναι κατά λέξη τα λόγια που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σημειώνω ότι χρησιμοποιεί τον όρο όχι κατάλληλη ή ε, επαρκή, αλλά ισοδύναμη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται λοιπόν ισοδύναμη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να προβούμε σε ανταλλαγή πληροφοριών με οδήποτε τρίτο κράτο, όπω ε, φερειπίνει Ηνωμένε ΗΠΑ. Τι στοιχεία είναι αυτά τα οποία χρειάζονται τώρα για να ε, στοιχειοθετηθεί ισοδύναμη προστασία και από τι δύο χθε του Ατλαντικού. Πρώτο στοιχείο. πρέπει να υπάρξει ως προϋπόθεση για την προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και μια σχετική ε, τακτική συνεργασία με τα μεταλλαγή πληροφοριών. Πρέπει λοιπόν και οι δύο εταίροι, ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπω αυτά αναγνωρίζονται και θεμελιώνονται μέσα από τι διεθνεί συμφωνίε και συμβάσει, το Διεθνέ Σύμφωνο για τι Πολιτικέ Ελευθερίε και τα Αστικά Δικαιώματα, το πρώτο προαιρετικό πρωτόκολλο την Αμερικανική Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Οικουμενική Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουν κυρώσει οι Ηνωμένε Πολιτείε για να μπορεί κανεί να προσφύγει ενώπιον των δικαστηρίων του, πράγμα το οποίο ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Όσο λοιπόν δεν ισχύουν αυτέ οι συμβάσει και δεν μπορεί κανεί να τι ε, επικαλεστεί ενώπιον ενό Αμερικανικού δικαστηρίου, υπάρχει ο κίνδυνο σε περίπτωση που διαθέτεται στοιχεία και προκύψει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο θυγόμενος, το θύμα, να μην μπορεί να προσφύγει στα Αμερικανικά δικαστήρια. Και δεν αρκεί, πιστεύω, το να εισάγεται σε μια διεθνή συμφωνία ρήτρα η οποία ε, θα επισημαίνει ότι δεν διατηθείται δεδομένα εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι κάθε ανταλλαγή στοιχείων σημαίνει και τον κίνδυνο της κατάχρησης των πληροφοριών που θα οδηγούσε ενδεχομένως σε παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Επομένως χρειάζεται να υπάρχει ένα ουσιαστικό πλαίσιο, ένα περιβάλλον κατάλληλο για την διαφύλαξη των ανθρωπινών δικαιωμάτων όπως αυτά εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, ένα άλλο στοιχείο που απαιτείται είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, των θεμελιώδες δηλαδή δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο και εδώ έχουμε να κάνουμε με εγγύσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα όσα περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαιτούνται δηλαδή πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την διαβίβαση και την χρήση προσωπικών δεδομένων από οποιονδήποτε εκ των εταίρων, πράγμα το οποίο συνεπάγεται ουσιαστικά με το να πούμε ότι δεδομένα που ε, διατίθεται σε περίπτωση ποινικών ε, διαδικασιών, διατίθεται μόνο εφόσον υπάρχει ουσιαστική και πραγματική υποψία περί διάπραξης αδικήματος, ότι τα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ε, ότι απαλήφονται αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν χρειάζεται η φύλαξη τους περαιτέρω για, ε, ότι δηλαδή έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχουν διατεθεί. Αυτό είναι κάτι στο οποίο επιμένουμε πάντοτε και ορίζει και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, δηλαδή πρέπει να απαλήφονται αμέσω τα δεδομένα, δεν μπορεί κανεί να τα φυλάσει για περιόριστο χρονικό διάστημα και αυτή η υποχρέωση πρέπει να είναι δεσμευτική. Επίση, ο λόγο για τον οποίο διατίθεται τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν δηλαδή πληροφορίε μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχουν ζητηθεί και διατεθεί. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Δεν θα μπορούν οι Αμερικανοί να χρησιμοποιούν δεδομένα ε, για για λόγο των οποίων δεν είχαν περιγράψει το αίτημα διάθεσης. Κάτι το οποίο, επί παραδείγματι, ιδιαίτερα υπογραμμίζουν ορισμένα ευρωπαϊκά δικαστήρια, όπως το, Ευρωπαϊκό, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Σταγματικό Δικαστήριο, τον ε, περιορισμό δηλαδή του, στόχου, σκοπού μάλλον χρήσης ε, των δεδομένων. Η άμεση ε, κοινοποίηση επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτή θα πρέπει να σωματωθεί στην διαπραγματευτική εντολή. Ένα τρίτο στοιχείο τώρα, πολύ σημαντικό, είναι η συνολική δυνατότητα ε, αποκατάστασης των δικαιωμάτων από τα δικαστήρια. Δηλαδή, η οσδήποτε θεωρεί θυχής ως προς τα δικαιώματά του θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφύγει στα δικαστήρια. Ε, το σχέδιο της συμφωνίας φαίνεται κάπως ασαφές γιατί λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της αποκατάστασης των δικαιωμάτων χωρίς όμως να ορίζεται συγκεκριμένα ποια είναι αυτή. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της ανεξάρτητης εποπτείας της προστασίας αυτών των δικαιωμάτων, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πράγμα που και πάλι είναι ασαφές διότι δεν, είναι, δεν υπάρχει επαρκής περιγραφή και ισοδύναμη περιγραφή αυτής της εποπτείας. Έτσι λοιπόν συστήνουμε τα εξής πρέπει να υπάρξει ως προϋπόθεση ισοδυναμή προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων προκειμένου να διατεθούν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Δεύτερον, θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκή και ισοδύναμα επίπεδα προστασίας των δεδομένων. Και τρίτον, θα πρέπει να δημιουργηθεί και, και ισοδύναμος δικαστικός ή δικαιικός μηχανισμός. Ε, και εδώ έρχομαι σε μία απόφαση του Γερμανικού Δικαστηρίου σε σχέση με την, κύρωση της ε, σύμβασης για την ε, ε, αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος, το οποίο γερμανικό δικαστήριο απεφάνθη ότι εφόσον δεν υπάρχει ισοδύναμη προστασία, δεν ισχύει η συμφωνία. Και αυτό είναι ο κίνδυνος που διατρέχουμε εάν δεν υπάρξει εξασφάλιση επαρκούς και ισοδύναμης προστασίας των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα το προηγούμενο τμήμα μας ήταν πιο πολιτικό. Το τωρινό εστιάζεται περισσότερο στις νομικές πτυχές. Τώρα θέλω να είμαι πολύ προσεκτική βέβαια στη διατύπωσή μου. Αναρωτιέμαι κατά πόσο όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ληφθεί επαρκώ υπόψη από την Επιτροπή και το Συμβούλιο και κατά πόσο στο τέλος της διαδικασίας θα μπορούν να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία η οποία να μπορέσει να αποδειχθεί επιτυχής μετά από τις δοκιμασίες που, στις οποίες θα την υποβάλουμε. Οι ειδικοί θα την υποβάλουν. Θα δώσω το λόγο στους συζητητές και μετά θα ζητήσω από τους συναδέρφους να μας πούν αν έχουν να κάνουν σχόλια. Ο εισηγητής. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τα όσα μας είπαν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι τα νομικά ζητήματα που προέρχονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αποσαφινιστούν. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για το θέμα PNR, υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια δεδομένα και το συνταγματικό πλαίσιο μερικές φορές είναι πολύ στενό όσον αφορά τη χρήση τους. Ή για να τα αποθηκεύσει κανείς. Το αφήνω εκεί. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές, ας προχωρήσουμε. Ωραία λέει Πρόεδρος. Οι συνάδελφοι τώρα έχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Από τόσο ακούσαμε, λέει ο κύριος Σταβάρης, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε σε τέτοιες συμφωνίες. Το θέμα είναι τι έχουμε πάρει, γιατί από τους ομιλητές που ακούσαμε ξέρουμε τι θέλουμε. Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια τέτοια συμφωνία. Αν είχαμε ξεκινήσει από αυτή τη βάση, δεν θα συζητάγαμε αυτά τα προβλήματα σήμερα. Οπότε ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Δεν έχω ερωτήσεις. Ο κύριος Μπρόντς, πολύ σύντομα. Ο κύριος Στεκλέρ είπε, αν το κατάλαβα καλά, ότι υπάρχει ήδη ένα σχέδιο συμφωνίας το οποίο θα συζητήσει το Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Εμείς έχουμε πρόσβαση σε αυτό. είναι η εντολή. Φυσικά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, λέει η Πρόεδρος. Όπως είπα και πριν, τα τελευταία τρία χρόνια οι υπηρεσίε τη Επιτροπής διαπραγματεύονται με τις Ηνωμένε Πολιτείε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμαρτυρήθηκε, διότι δεν είναι ένα καθαρά διοικητικό θέμα. Αλλά βέβαια είχαν προχωρήσει ήδη πολύ. Μόνο ένα-δύο θέματα έμεναν. Τώρα υπάρχει ένα σχέδιο εντολής Φαντάζομαι ότι μπορεί κανείς να το δει. Μπορούμε να το δούμε σε secure room. Αλλά όχι να το συζητήσουμε. Που νομίζω ότι είναι γελίο, γιατί στο κάτω-κάτω πρόκειται για τα δεδομένα των πολιτών μας. Αν οι πολίτες μας πρέπει να υποβάλουν όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, εάν μη τι άλλο θα πρέπει και εμείς να τους προσφέρουμε το ίδιο επίπεδο πρόσβασης στις διαπραγματεύσεις γι' αυτά. Έχω και άλλη μια ερώτηση, λέει ο κύριος Μπρόνς. Υπάρχουν δύο δυνατότητες. Η μία είναι η νέα αυτή συμφωνία να είναι συμπληρωματική επί της διαδικασίας. Αλλά μπορεί η νέα αυτή συμφωνία να είναι μια πλήρης νέα ουσιαστική συμφωνία που να καλύπτει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες. Τι από τα δύο. Αυτό θα συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση, αλλά είχε συζητηθεί λιγάκι και στην ε, στο πρώτο μέρος για το κατά πόσο αναδρομικά ή όχι θα ισχύσει. Αλλά πρέπει να διευκρινιστεί ακόμα, συμφωνώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Η συμφωνία αυτή που τώρα βλέπουμε σαν συμφωνία πλαίσιο δεν πρέπει και δεν θα είναι η βάση για την μεταφορά δεδομένων και για την ανταλλαγή δεδομένων. Κάθε φορά θα υπάρχουν ειδικέ συμφωνίες που θα ρυθμίζουν για ποια δεδομένα μιλάμε, ποια μεταβιβάζονται και ποια δεν μεταβιβάζονται. Θα αποτελεί όμως μια συμφωνία πλαίσιο, ομπρέλα, που θα θέτει τις αρχές της συμφωνίας και θα βασίζεται στις γενικές αρχές της προστασίας δεδομένων. Το ζήτημα για μας τώρα είναι κατά πόσο θα πρόκειται για μια πλήρη προσέγγιση από πλευράς Ευρώπης, ώστε να καλύπτουμε όλες τις συμφωνίες μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πάντως δεν αντικαθιστά τις συμφωνίες αυτές. Τις πλαισιώνει. Να προσθέσω κι εγώ δύο λόγια σε αυτό. Οι ειδικέ συμφωνίες χρειάζονται έτσι ώστε μιλάμε για τα σωστά δεδομένα και δεν προσθέτουμε κι άλλα που δεν θα έπρεπε στην ε, συμφωνία αυτή. Λέει η κυρία Γκαρέλ. Πρόεδρος, δεν έχει γίνει ακόμα όμως η δοκιμασία, έτσι δεν είναι όσον αφορά τα PNR. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. Παρακαλώ, μήπως θέλετε κι εσείς να απαντήσετε. Χαίρομαι που ακούω και εγώ ότι η συμφωνία αυτή δεν έχει σαν σκοπό πιο ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Δεν ήταν σαφές πριν αυτό. Βέβαια είναι απογοητευτικό που δεν έχουμε περισσότερη πρόσβαση στα σχέδια γράφων και γενικά στα έγγραφα που συζητιούνται. Διότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε κι εμεί να έχουμε επικοδηματικά σχόλια άμα δεν ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και για εμά του ερευνητέ, ε, του μελετητέ, του αναλυτέ που παρακολουθούμε στενά αυτά τα ζήματα, 12-14 ε, σελίδε για ένα τέτοιο θέμα δεν είναι τίποτα. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να μπορούμε να πούμε και εμείς την απόψή μας. Ναι, συμφωνώ λέει ο Πρόεδρος θα ερευνήσουμε περισσότερο ποιοι είναι οι κανόνες για την πρόσβαση σε τέτοιου είδους έγγραφα. Συχνά όταν κάνουμε διαπραγματεύσεις για οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία, είναι η άλλη πλευρά που ζητάει να μείνουν απόρριτα κάποια έγγραφα. Και τότε τι γίνεται, οι δικές μας οι προδιαγραφές δεν ισχύουν πια. Τι τις έχουμε τις δικές μας τις προδιαγραφές. Και πάλι εδώ δεν μιλάμε για τεχνικά ζητήματα, μιλάμε για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών μας. Έχουν το δικαίωμα να ξέρουν και εμείς ως Κοινοβούλιο πώς θα ελέγξουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές αν δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να συζητάμε μεταξύ μας τα έγγραφα τα οποία συζητιούνται στις διαπραγματεύσεις. Ε, από ό,τι όμως έμαθα ήδη έχει δημοσιευθεί κάτι στο Stakewatch, τουλάχιστον εκεί κάτι μπορούμε να βρούμε. Ωραία, τελειώνουμε και με αυτό το μέρος και περνάμε στο τρίτο και τελευταίο. Α, κύριε Μπρέγερ, μήπως εσείς έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις. Μια που δεν συζητήσαμε αρκετά την σχέση των ε, προηγούμενων συμφωνιών και της τωρινής, επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποια σχόλια, λέει ο κύριος Μπρέγερ. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει μια μήνυμου προδιαγραφή. Να δούμε από εκεί και πέρα ειδικέ συμφωνίες τι μπορούν να προσθέσουν για την μεταφορά, για παράδειγμα, δεδομένων που πρέπει να είναι πιο αυστηρά από μια άποψη, αλλά από την άλλη μελευρά μπορεί να είναι ε, ευρύτερε οι προδιαγραφέ. Η νέα συμφωνία μπορεί να θέσει τα νέα, τη νέα βάση για το επίπεδο προστασίας. Μερικές φορές χρειάζονται υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Πρόεδρος, ναι, αυτή είναι και η πρόθεση. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Τι σημειώσεις που έχετε για τις παρεμβάσεις σας αφήστε τες στην γραμματεία αν δεν σας πειράζει για να τις έχουμε. Και περνάμε, λάμε, ε, περνάμε λοιπόν στο τρίτο μέρος, στο τρίτο πάνελ. Uh, λοιπόν, συνάδελφοι, το τελευταίο και τελικό θέμα για σήμερα που αφορά τις ε, επιπτώσεις της νέας συμφωνίας πλαίσιο στις διμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολυμερείς σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους ομιλητές να μην ξεπεράσουν τα 10 λεπτά ο καθένας. Δεν θα σας ενοχλήσω μέχρι τα 10 λεπτά και μετά θα υπάρξουν ερωτά απαντήσεις. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Τρολ Σόρτινγκ, βοηθός διευθυντής της Ευρωπόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να επιταχύνω τη συζήτηση. Η συνεργασία ΕΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό μπορεί να γίνει με θεσμικό τρόπο και με πολλές μορφές. Υπάρχουν αξιωματικοί σύνδεσμοι που συναντώνται στο κτίριό μας στη Χάγη, στα πλαίσια της Ευρωπόλ, όπως επίσης και δύο αξιωματούχοι της Ευρωπόλ στην Αμερικανική πρωτεύουσα, όπου έρχονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και τους ομολόγους τους. Έχουμε επαφές και με το ATF, ε το FBI, την Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Προστασίας Συνόρων και την Ταχυδρομική Υπηρεσία της Αμερικανικής Κυβέρνησης και υπάρχουν 27, 23 θέματα μάλλον στα οποία προσπαθούμε να κινητοποιηθούμε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα Έχουμε αρκετές περιπτώσεις τις οποίες έχουμε βοηθήσει να διαλευκάνουμε, ιδιαίτερα στη σεξουαλική κακομεταχείριση των παιδιών. Έχουμε ενημερώσει τις Ηνωμένε Πολιτείες, περιπτώσεις τις οποίες οι ίδιοι Αμερικανοί δεν γνώρισαν. Εμείς έχουμε το δίκτυο CN, Λέγεται Σιένα το σύστημά μας, χρησιμοποιείται αποκλειστικά φυσικά από την Ευρωπόλου και έχει σαν στόχο την προστασία της εμπιστευτικότητας και χρησιμοποιούμε δικτυακές ρυθμίσεις ιδιαίτερως απαραβίαστες και ασφαλείς. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν και τις ελλείψεις που έχουν σημειωθεί. Οι εμπειρίες μας μας δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΙΠΑ έχουν κοινά χαρακτηριστικά στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά υπάρχουν επίσης και πολλές διαφορές. Σαν παράδειγμα, πολλά θέματα τα οποία ρυθμίζονται στα πλαίσια της νομικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιμετωπίζονται πάρα πολύ πιο θεωρητικά από τις αμερικανικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Γι' αυτό η νέα αυτή συμφωνία πλαίσιο θα πρέπει να βοηθήσει να ενισχύσει την συνεργασία μας σεβόμενη πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στην Ευρωπόλ έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα αυστερό προστασία των δεδομένων. Είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα στο σύνολο των αστυνομικών δυνάμεων και στην Ευρώπη και τα συστήματά μας τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από άλλες δυνάμεις αντίστοιχες στον κόσμο. Το θέμα είναι πώς η νέα συμφωνία μπορεί να επηρεάσει τις ισχύουσες συμφωνίες με, την, ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείες για την τροφοδοσία σε στοιχεία της Ευρωπόλ. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας νέας προοπτικής αξιολογώντας τους μηχανισμούς ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Βασική μας ανησυχία είναι ότι η Ευρωπόλ θα πρέπει να ενισχύσει ακόμα υψηλότερα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και αυτό θα ρυθμίζεται από την ε, συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Το θέμα είναι λοιπόν αν θα πρέπει η νέα συμφωνία να ισχύει για τις μελλοντικές ρυθμίσεις που θα γίνουν ή αναδρομικά και για τις ρυθμίσεις που έχουν αποφασιστεί μέχρι τώρα. Κάποιοι εμπλεκόμενοι πιστεύουν ότι η συμπερίληψη των ισχυουσών συμφωνιών είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Πιστεύουν ότι αυτές οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι δεσμευτικές για τις μελλοντικές μόνο συμφωνίες. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Ε, οργανώσεις όπως η Europol και η Eurojust στην ουσία θα αγνοηθούν αν υπάρχουν ε, περίπλοκες ε, πλέον ρυθμίσεις με τη ΣΥΠΑ. Ο κίνδυνος είναι η Ευρωπόλ να αγνοηθεί γιατί τα κράτη-μέλη θα βλέπουν την συνεργασία με τη ΣΥΠΑ μέσω ημών σαν ένα επιβαρυντικό ουσιαστικά στοιχείο και ε, κάτι το οποίο θα καθιστά τις συμφωνίες λιγότερο αποτελεσματικές. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ε, να συνεχίσουμε να βοηθάμε τους Ευρωπαίους πολίτες στα πλαίσια ενός ε, πλαισίου το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των ανταλλαγών στοιχείων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και, της, ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως της νομικής βάσης. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ταυτόχρονα είναι και προς το συμφέρον της κοινότητας της αστυνομικής έτσι ώστε τα ίδια επίπεδα προστασίας να εφαρμόζονται σε όλες τις πλευρές. Αυτά τα στοιχεία, εφόσον είναι συνεκτικά, είναι υψηλού επίπεδου, έχουν υψηλή ακρίβεια και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Αυτό είναι σημαντικό και για την Ευρωπόλ, αλλά και για όλες τις διμερείς μορφές συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Για να κλείσω, επιστρέψτε μου να πω ότι η αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ζωτική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και των σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε αποτελεσματικές λύσεις προώθησης της διατλαντικής συνεργασίας σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπόλ είναι ολόψυχα αφιερωμένη την προστασία των υψηλών επιπέδων προστασίας με τη σειρά τους των προσωπικών δεδομένων και αναγνωρίζουμε βέβαια ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να επηρεάσει την συνεργασία μας με τη ΣΥΠΑ. Παρ' όλα αυτά εμείς θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα θέματα στα οποία, για τα οποία καλούμεθα να είμαστε αποτελεσματικοί και θα συνεργαστούμε μαζί σας όποτε το επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν πολύ σύντομος. Έχουμε δημιουργήσει παράδοση έτσι ώστε να μην ξεπερνάει κανείς τον χρόνο του. Η κυρία Γκαμπριέλ Τσίτς έχει το λόγο. Είναι μέλος της Βουλής της Σλοβενίας και πρόεδρος της ομάδας εξωτερικών σχέσεων του Eurojust. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ε, πρόσκληση που απευθύνατε στην Eurojust ε, να συμμετάσχει στην ακρόαση σας σήμερα. Πρόκειται για μια ευπρόσδεκτη ευκαιρία να συστήσουμε θέματα πολύ σοβαρά και γνωρίζουμε βεβαίω ότι είναι ύψη τη σημασία για όλου μα τα θέματα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Eurojust έχει αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή μια συμφωνία συνεργασία με τι ΗΠΑ τη Αμερική που συνήθισε στι 6 Νοεμβρίου του 2006. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ε, περιέχει σημαντικές και εκτεταμένες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συγκεκριμένα 23 πρόνοιες, δηλαδή άρθρα, του, της συμφωνίας και συγκεκριμένα τα άρθρα 8-19 της συμφωνίας ε, ασχολούνται ιδιαίτερα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. δεδομένων. Και έτσι προσφέρουν μια εκτεταμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα να σας δώσω συγκεκριμένες πληροφορίες ως προς το τι καλύπτεται σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή υπάρχει η άδεια για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο περιορισμός της χρήσεως προσωπικών και λοιπόν δεδομένων, διαβίβαση ορισμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, η προστασία, η διαφύλαξη, η διαφάνεια, η ασφάλεια, η πρόσβαση, η διόρθωση και ε, παρεμπόδιση διόρθωσης, ο περιορισμός ο χρονικός ε, και της χρήσης, η επισκόπηση της ε, χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Αυτά ορίζει η ίδια συμφωνία που έχουμε με τις Η συμφωνία λειτουργεί ομαλά ικανοποιητικά και εφαρμόζεται ικανοποιητικά και από τις δύο όχθες του αθλητικού. Υπό αυτό το, το φως αυτό των εξελίξεων λοιπόν θεωρούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την υφισταμένη κατάσταση. Τούτου λεχθέντος όμως η Eurojust διατηρεί ανοιχτή την προοπτική και τη διάθεση να συζητήσει και να συνομιλήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη αυτής της ενδιαφέρουσας πρωτοβουλίας. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω ότι θα ήθελε η Eurojust ε, να εξασφαλίσει ε, ευθυγράμμιση της συνεργασίας που έχει αυτή τη στιγμή με τις ΗΠΑ με ένα νέο πιθανό ε, σύνολο συμφωνιών εφόσον υπάρχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων από αυτό που προκύπτει από την υφισταμένη συμφωνία. Και πάλι στο ίδιο πνεύμα και με στόχο την διαφύλαξη του υφισταμένου επίπεδου προστασίας. Ελπίζουμε ότι μια μελλοντική συμφωνία πλαίσιο θα περιλαμβάνει και ρήτρα που θα υποδεικνύει πως το φυστάμενο επίπεδο προστασίας ήδη συνηθισών συμφωνιών θα διαφυλάσσεται κατά πάση περιπτώση. Εν πάση περιπτώσει. Πλην όμως αναγνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερο σχέση με την υφιστάμενη συμφωνία πλαίσιο και ενδεχόμενε συμφωνίες που υπάρχουν όπως το πλαίσιο της ειδικέ συμφωνίες δηλαδή προς το πλαίσιο της Eurojust ε, έχουμε ε, να κάνουμε πολλά λεπτά ευαίσθητα και επικίνδυνα νομικά ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν ε, και να αντιμετωπιστούν σωστά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ο χώρο στον οποίο κινείται και λειτουργεί η Eurojust. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία το να βεβαιωνόμαστε σε κάθε περίπτωση ότι δεν διαταράσσεται η ασφάλεια δικαίου στου ε, τομεί αυτού και ότι οι πιθανέ ε, συλλήψει ή και καταδίκε που έχουν ενδεχομένω λάβει χώρα ε, ή υπ' αυτό το καθεστώ δεν θα οδηγήσουν σε κίνδυνο για δικαστικές αγωγές ή άλλους αγώνες ή προσβολές κατά την περίοδο αυτή με τη νέα περίοδο. Η συνεργασία λοιπόν με, ε, θεσμικά, με οργανώσεις όπως η Eurojust θα πρέπει να υποταχθεί στις νέες συνθήκες εφόσον υπάρξουν, νέες συμφωνίες δηλαδή, ή εφόσον το ε, ακολουθούν την εφαρμογή προηγουμένων συμφωνιών και τα άλλα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αδίποτε λύσεις δοθεί θα πρέπει να ισχύει ισοδύναμα και για τα κράτη-μέλη και για τις ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες για την ε, εφαρμογή επιβολή του δικαίου ε, ιδάλλως κινδυνεύει να διαταραχθεί σημαντικά η συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η Eurojust, θα θέλω να υπογραμμίσω, με πολύ μεγάλη χαρά θα συνεχίσει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πολύ λεπτό και ευαίσθητο αυτό θέμα, προκειμένου να εξασφαλίσει πώς η κατάσταση, όπως θα εξελιχθεί στο μέλλον και ανεξαρτήτως ε, της ιασδήποτε ε, νομικής λύσης που θα προκύψει, θα είναι προ το συμφέρον τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων και του ιδιωτικού βίου των πολιτών μα. Και για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία που δώσατε να εκφράσουμε τι θέσει τη Eurojust στη συνεδρίαση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Με χαρά ακούω ότι και η Europol και η Eurojust υποστηρίζουν την ιδέα την πρόθεση να υπάρχει ένα στο επίπεδο προστασία από τι δύο πλευρέ. Ο κύριο Μιχαήλ Χάιν τώρα. Χάιν ή Χάιν επικεφαλής της Μονάδας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στο μέα της αστυνομικής συνεργασίας, της αστυνομίας, ε, της καταπολέμησης της εγκληματικότητας στη Γερμανία. Μια, μέσα σε μια υπηρεσία η οποία γνωρίζουμε ότι διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστώ για την πρόσκληση τη δική σας, των συναδέλφων σας από την Επιτροπή των ε, Πολιτικών Ελευθεριών ε, να συμμετάσχουμε σε αυτή τη ε, διάσκεψη και να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Σάου, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει λόγω της υποχρέωσης του να παρασύρει μια πολύ σημαντική διάσκεψη στην Ιερουσαλήμ για το ίδιο θέμα. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν και τον αντικαθιστώ εγώ. Θα ήθελα να πω το εξή. Ο Γερμανός διαμεσολαβητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, καλωσορίζει την ε, πρόταση για μια δεσμευτική σειρά ε, προστασίας, μέτρων προστασία των προσωπικών δεδομένων σε μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό με την ελπίδα ότι θα εξασφαλιστεί σε επίπεδο τόσο Ηνωμένων Πολιτειών όσο και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη νέα αυτή συμφωνία μια σειρά δεσμεύσεων για υψηλό επίπεδο κατά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό λοιπόν το έχουμε υπογραμμίσει και σε μια προηγούμενη αρχές του έτους διάσκεψη των αρχών εποπτείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια σειρά προτάσεων, ιδιαίτερα στο άρθρο 29 της ανακοινωσής μας, μια διάσκεψη στην οποία έλαβε μέρος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά την οποία εμείς χαιρετήσαμε την πρόταση για νέα συμφωνία. Όσον αφορά τώρα τη σχέση της, ε, της νέας συμφωνίας με τις υφιστάμενες, θα ήθελα να κάνω την εξή παρατήρηση. Η ΥΠΑΤΗ Αρχή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία θεωρεί ότι η οδήποτε νέα συμφωνία θα πρέπει να ισχύσει και στι υφιστάμενε συμφωνίε και σε ιεσδήποτε ενδεχόμενε διμερεί συμφωνίες έχουν συναυθεί μεταξύ ΗΠΑ και κρατών μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Υπάρχει μια εξέλιξη διμερών συμφωνιών συγκεκριμένα, ε, είτε επίκαιρη είτε ε, προβλεπόμενη στο άμεση μέλλον, ε, συμφωνιών που ονομάζονται Prim-like και η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση από πλευρά των αρχών της μίας της άλλης πλευράς σε δεδομένα όπως δακτυλικά αποτυπώματα, προσωπικά στοιχεία, και με στόχο την ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και τη διεθνούς τρομοκρατία. Οι αρχέ προστασία των προσωπικών δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνουν ότι αυτέ οι συμβάσει, οι διμερεί, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασία των προσωπικών δεδομένων και ω εκ τούτου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντίστοιχε αρχέ, να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασία. Πράγμα το οποίο θα οδηγούσε όχι μόνο σε βελτίωση του επίπεδου προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα και σε μια ενίσχυση τη εναρμόνιση αυτών των προσωπικών δεδομένων, τη προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Με τη συμφωνία αυτή, τουλάχιστον αυτό ισχύει όσον αφορά τη συμφωνία που έχει συνάψει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία με τι ΗΠΑ, προβλέπεται ότι προβλέπονται κάποιες αρχές οι οποίες υπολείπονται των όσων έχουν ε, διατυπωθεί ως βασικές αρχές από την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας ε, Προσωπικών Δεδομένων. Με αποτέλεσμα τα κενά αυτά που προκύπτουν από τις ε, εν λόγω διμερείς συμφωνίες να σημαίνουν πως χρειάζεται να συμπληρωθούν, να καλυφθούν με νέες διαπραγματεύσεις, νέες συμφωνίες. Επίσης, μεταξύ Γερμανίας και ε, ΗΠΑ Αμερικής υφίστανται τέτοιες συμφωνίες, όπως μια η οποία συνήθι το 2002, και η οποία δεν μπόρεσε να κυρωθεί λόγω των δεσμεύσεων ε, και του χαρακτήρα του Ομοσπονδιακού της Γερμανίας, γιατί ένα από τα κρατήδια του Ομοσπονδιακά αρνήθηκε την κύρωση, ως αρχή αρμόδια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, Επισημαίνουμε επίσης μια σειρά από ελλείψεις ε, σε σχέση με την υφιστάμενη διμερή συμφωνία της ε, Γερμανίας με τις ΗΠΑ που θα μπορούσαν οι ελλείψεις αυτές να ε, διασκεδαστούν, να διευθετηθούν εφόσον υιοθετηθεί μια νέα συνολική συμφωνία. Ελλείψεις και κενά σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής ενός ιδιώτη ή ε, της ε, εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων από τη μία χώρα στην άλλη. Τέτοια στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να προκύψουν μέσα από μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία και να ε, ρυθμίσουν τα κενά κατά τρόπον ώστε, που η, κατά τρόπον ώστε η, η σύμβαση, η συμφωνία η οποία θα κυρωθεί να ισχύει δεσμευτικά και στις ΗΠΑ όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν ε, πιστεύουμε ότι η εντολή που θα προσδοριστεί για τη διαπραγμάτευση θα πρέπει να ορίζει και ε, ρήτρε επανεξέταση με συγκεκριμένε προθυσμίε ώστε να επιβεβαιώνεται ότι έχουν όντω καλυφθεί τα νομοθετικά κενά, τα κενά στην νομοθεσία. και πιστεύουμε ότι θα πρέπει μια νέα συμφωνία να προβλέπει αυστηρέ διατάξει προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η αρχή, την οποία εκπροσωπώ επίση, ε, πιστεύει ότι θα πρέπει να καλύπτονται από μια νέα συμφωνία ε, και άλλες ενδεχομένως η PNR, η SWIFT συμφωνίες τομεακές δηλαδή, συμφωνίες που έχουν να κάνουν και με την συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως αεροπορικές εταιρείες κτλ. ή με κρατικές υπηρεσίες και αρχές των ΗΠΑ. Σε σχέση λοιπόν με το άρθρο 29 και τη σχετική ομάδα που το προσυπέγραψε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η εξέλιξη και σημειώνουμε ότι παρά τις κάποιες επικρίσεις ως προς την συμφωνία SWIFT και την PNR, θεωρούμε ότι αυτές οι συμφωνίες παρεμβαίνουν και παραβιάζουν πολλά δικαιώματα αθώων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μια κάποια αποτελεσματικότητά τους και θα πρέπει να ε, καλυφθούν από μια νέα συνολική συμφωνία ώστε να καλυφθεί το κενό ε, στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Η τελευταία σα παρατήρηση για την συμφωνία PNR ε, θα ήθελα να πατήσω εδώ ότι δεν έχει συναυθεί ακόμα αυτή η συμφωνία και σε δεν ξέρουμε τι μορφή θα λάβει. Για το άλλο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο είναι αλληλεύεται ασφαλώ, για τις διμερεί ε, συμφωνίε λεγόμενε ε, prim -like, και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που κάνατε εσεί την παρατήρηση. Κατά τα άλλα, όμω, δεν είμαι και τόσο ικανοποιημένη για το γεγονό ότι ομόλογοι από άλλα κράτη-μέλη δυστυχώ δεν είδαν την ίδια αναλογία, γιατί βλέπουμε ότι πολλέ είναι οι διμερεί συμφωνίε που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και ΗΠΑ, πολλέ δε φορέ χωρί καν να υποβληθούν προσκύρωση στα εθνικά κοινοβούλια. Και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι ιδιαίτερω για την ε, για τι αρμοδιότητε και την δραστηριότητα που επιδεικνύει η αρχή, η πατριαρχή για την προσοχή των προσωπικών δεδομένων τη Γερμανία. Ε, ο επόμενο ομιλητή. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντόουε Κόρφ, ε, Ολλανδός φυσικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λέει Ολλανδικά πρώτα ο κύριος Κόρφ. Και συνεχίζει αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή που με κάλεσε να έρθω εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσω σύντομα να σας παρουσιάσω τα θέματα μου, αλλά πριν μπω στα ειδικά θέματα θα ξεκινήσουμε κάποια γενικά. Η παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη σήμερα νωρίς το απόγευμα ήταν πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, από τη μια μεριά μιλάει για κοινέ αξίες, για τον πυλοφράτη των Ηνωμένων Πολιτειών, που αποτελεί τη βάση για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αμερική και στην Ευρώπη. Βέβαια έχουν ε, προδοθεί αρκετές από αυτές τις αξίες, όπως είπε και ο Πάτρικ. Βλέπουμε να γίνονται παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων και βασικών δικαιωμάτων από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό και ήταν κάπως απογοητευτική ε, η παρέμβαση αυτή, διότι τελικά τα συνταγματικά δικαιώματα είναι περιορισμένα σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με μη Αμερικανούς πολίτες είτε στο Γουαντάναμο είτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και δεν μπορούμε εμείς να αποστασιοποιηθούμε. Από την άλλη μεριά βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να προσφέρει καλή νομική προστασία. Άρα είναι θέμα του πώς αντιλαμβάνεται κανείς την ε, επικοινωνία. Σίγουρα η κυβέρνηση Μπούς υπονόμευσε πολύ την κατάσταση γιατί αγνόησε τους κανόνες. Η Αμερική λοιπόν μπορεί να κάνει πολλά, αλλά πρέπει να δεχτεί να συνεργαστεί με την Ευρώπη. Τώρα ας μπούμε στο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Και πάλι ο πρέσβης είπε ότι έχουμε κοινέ αξίες, κοινέ αρχές, αλλά έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Μα ακριβώς αυτό είναι και το ζήτημα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα στις Ηνωμένε Πολιτείες που να είναι κοντά στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων ή που να μοιάζει με αυτά που προσπαθεί να πετύχει η Ευρώπη ή η Γερμανία για αυτό το θέμα. Έκανα μια μεγάλη μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις νέες προκλήσεις στο θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ε, φαντάζομαι να ενημερωθείτε κι εσείς. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και η μελέτη του καθηγητή από το Berkeley, του Μάρκιν, που αναφέρεται στην προστασία δεδομένων στι Ηνωμένες Πολιτείες. Και από εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι τα κενά και πού δεν τηρείται η προστασία προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως το ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί και αυτό είναι πολύ βασικό. Και είναι αυτό το οποίο θέλουμε εμεί οπωσδήποτε. Γιατί δεν μπορεί να έχει ένα καθεστώ προστασία ε, δεδομένων αν χρησιμοποιεί την έννοια τη συνήθω χρήση. Αυτό κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, που εμεί δεν το θέλουμε. Ούτε μπορεί να έχει ένα σύστημα χωρί ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Το χρειάζεται κανείς. Δεν μπορείς να έχεις προστασία δεδομένων ούτε μπορείς να ακούς οι Ηνωμένες Πολιτείες να λένε εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε τις αρχές της Privacy Act, του νόμου δηλαδή για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Αλλά εκεί υπάρχουν τόσα πολλά κενά και τόσες πολλές ελλείψεις που τελικά δεν γίνεται να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει δικαίωμα στην πρόσβαση, δεν υπάρχει δικαίωμα στη διόρθωση, σε αλλαγές των δεδομένων αυτά. Κάπου αλλού για τις πανικές αρχές έχω περιγράψει, σε άλλο αγγραφό μου δηλαδή, πόσο, ανόητο, πόσο ανόητη είναι αυτή η προσέγγιση των ΗΠΑ και ότι έχουν συστήματα τα οποία δεν είναι κατανοητά. Ε, καθορίζουν ποιο είναι τρομοκράτη ανάλογα με τον τρόπο που περπατάνε, που στέκονται. Τους δεν μπορούμε εμεί να επιτρέψουμε δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών να συμπεριληφθούν σε τέτοια νόητα συστήματα. Δεν μπορεί να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτό, γιατί έπαξε και ένα δεδομένο μπει σε ένα σύστημα, υπάρχει στο σύστημα και τελείωσε. Δεν υπάρχουν μεταπεριορισμοί στις ΗΠΑ για τα δεδομένα αυτά. Ούτε ακόμα και για εκείνα τα οποία έχουν κάποιους περιορισμούς. Εκείνα που δεν έχουν, ξεχάστε το. Για πολλά χρόνια έχω δουλέψει στην κατάρτιση δικαστών, ερευνητών, στο Τουρκμενιστάν για παράδειγμα, όσον αφορά την χρήση βαναστηρίων. Και τους εξηγούσα ότι δεν μπορείτε να περιμένετε ε, καλή συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν εσεί χρησιμοποιείτε τα βασανιστήρια. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σα για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, αν χρησιμοποιείτε βασανιστήρια. Και εμεί λοιπόν το ίδιο πρέπει να πούμε στου Αμερικανού. Αν θέλετε να συνεργαστούμε μαζί σα, πρέπει να έχετε ένα σύστημα αξιοπρεπέ προστασία δεδομένων. Αλλιώ εσεί κάνετε αδύνατη την ε, συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο και όχι οι Ευρωπαίοι. Η επιστολή της Ένωσης Δικαιωμάτων των ε, Πολιτών έλεγε ακριβώς αυτά. Αντί να προσπαθούν οι Αμερικανοί να υποβιβάσουν, να χαμηλώσουν τις προδιαγραφές της Ευρώπης, πρέπει να κάνουν το αντίθετο, να ανυψώσουν τις δικές τους, όχι να δείχνουν τέτοια έλλειψη βούλησης. Ας περάσω λοιπόν τώρα στα ειδικά θέματα για το είδος της συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα έχετε δίκιο κυρία Πρόεδρε. είναι γελίο. Ναι, βλέπετε, εμείς λέμε πολλές φορές στην Αγγλία Mrs. Chairman, αλλά εγώ πώς να σας αποκαλέσω, Chairwoman. Πρέπει να δούμε τη συμφωνία άπαξ και έχουμε το κείμενο μπροστά μας. Και τότε να συζητηθεί ανοιχτά αυτό. Και στις διμερείς συμφωνίες είναι ενδιαφέρον που ακούσαμε τον πρέσβη να μιλάει και εκατοντάδες τέτοιες συμφωνίες. Εγώ μια-δυο έχω δει. Υπάρχει η Γερμανία-Αμερική συμφωνία. Το κοίταξα στο Eurostar σήμερα το πρωί στο τρένο και προσπάθησα να δω τις λεπτομέρειες. Ε, λοιπόν, υπάρχουν τόσα πολλά κενά. Οι ορισμοί δεν είναι σωστοί. Οι, τα πεδία εφαρμογή, τα δικαιώματα που αναφέρονται, υπάρχουν τόσα πολλά κενά που είναι λογικό να είμαστε επικριτικοί. Αν λοιπόν θέλουμε μια καλύτερη συμφωνία, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει, όπως είπε και η υποπτική αρχή, ένα πλαίσιο που να καθορίζει τις αρχές, το οποίο όμως δεν θα καλύπτει τα πάντα. Είναι σίγουρο. Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται στην ε, με ε, την κατασκοπία. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τα ίδια δεδομένα, αλλά χρησιμοποιούνται στην αστυνομική συνεργασία, στην επιβολή του νόμου. Μην προσπαθούμε όλα αυτά να τα καλύψουμε με μια συμφωνία πλαίσιο. Μπορείς να έχεις μια συμφωνία πλαίσιο που να αναφέρει τις αρχές, που να αναφέρει το πεδίο εφαρμογής και να λέμε ότι εφαρμόζεται στα κράτη, στην Αμερική, στην Ευρώπη, που ακόμα και αυτό ήταν δύσκολο. Οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να υποσχεθούν τίποτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, από εκεί και πέρα, πρέπει να υιοθετήσουμε πιο συγκεκριμένε συμφωνίε, όπω είναι το SWIFT, το PNR και όπω λένε και η Europol ε, και άλλοι, με τίποτα να μην κατέβουμε όσον αφορά το επίπεδο των προδιαγραφιών που θέλουμε για την προστασία. Να τηρήσουμε τα δικά μας επίπεδα προστασίας ή και παραπάνω. Με τίποτα να μην τα μειώσουμε. Πρέπει να επιμείνουμε όλες αυτές οι συμφωνίες να καλυφθούν. Και κάτι άλλο τώρα εμπόδιο που βάζει η Αμερική και ο πρέσβης, ο οποίος μιλάει για αναδρομική συμφωνία. Κανείς δεν το λέει αυτό. Κανείς δεν λέει ότι θα εφαρμόζεται η συμφωνία για πέντε χρόνια πριν τι έχει γίνει. Αυτό είναι ουσία, δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε να πούμε ότι άπαξ και η συμφωνία πλαίσιο έχει εγκριθεί, όλες οι σημερινές συμφωνίες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη νέα συμφωνία. Αυτό ναι, είναι φυσιολογικό. Εδώ δεν βλέπω τίποτα το περίεργο με αυτό. Μπορεί να χρειαστούν λίγα χρόνια. Θα γίνει. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πόσες είναι, εκατοντάδε είναι αυτές οι συμφωνίες. Πολύ θα ήθελα να τι δω. και πολλοί από εμά να ξέρετε, ευχαρίστω να καθίσουμε να τι μελετήσουμε και να σας πούμε τι στραβό έχει κάθε μία. Και να προσπαθήσουμε να τις διορθώσουμε λοιπόν μετά. Και να πούμε ότι οι συμφωνίε αυτές που ήδη υπάρχουν θα ισχύουν στο βαθμό που είναι συμβατές με την Γενική Συμφωνία Πλαίσιο. Είμαι κάπως απεσιόδοξος. Κάνω την Κασάνδρα εδώ. Και σα προειδοποιώ, όχι εσά το Κοινοβούλιο απαραίτητα, αλλά σίγουρα την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το εξή. Αν δεχτείτε μία συμφωνία η οποία αντιβαίνει στις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων της Ευρώπης, τότε ε, βάζετε σε κίνδυνο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάζετε το θεμελιώδη χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα έχετε και τεράστια προβλήματα, ενώ ήδη υπάρχουν όσον αφορά το, την αποθήκευση δεδομένων, με τα συνταγματικά δικαστήρια πολλών χωρών. Υπονομεύεται έτσι ολόκληρο το ευρωπαϊκό πλαίσιο και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί τα κράτη-μέλη και τα συνταγματικά δικαστήρια θα αρνηθούν να συμμορφωθούν με ε, συμφωνίες που δεν τηρούν τις προδιαγραφές που έχουμε τώρα. Ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν, θεμελιώδης χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευρωπαϊκά επίπεδα προστασίας. Αν οι Αμερικανοί συμφωνούν και θέλουν κάτι τέτοιο και μπορούν να το εφαρμόσουν εκεί, ευχαρίστως να συνεργαστούμε μαζί τους όπως μπορούμε. Αν δεν το κάνουν, τότε οι Αμερικανοί είναι εκείνοι οι οποίοι σαμποτάρουν το όλο εγχείρημα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπατε. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Να πω ότι ίσως είναι λάθος να λέμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν σέβονται τα επίπεδα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ νομίζω ότι με βάση τις εμπειρίες μας ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τα εκχωρούν όλα δεν πρέπει να κατηγορούμε τους Αμερικανούς, αυτοί ζητούν. Και αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ε, τα παραδίδουν, τότε υπάρχει ένα θέμα. Δεν μιλάω μόνο για το PNR, ξέρετε και το Ουσμπεκιστάν. Είχαμε επίσης μια έρευνα, επιτροπή έρευνας εδώ για τις παράνομες μεταφορές από τη CIA και ε, καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν έχει, ε, θα έλεγα, αξιολογηθεί σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό των Αμερικανών, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί. Ασκούμε κριτική στον Κουαντάναμο, αλλά δεν ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία βοήθησε να πάνε το 90% των ε, εγκλήστων στον Κουαντάναμο. Λοιπόν, δεν πρέπει να λέμε ότι είναι από τη μία η κακή και από την άλλη καλή Ευρωπαίοι. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρώτη προσωπική παρατήρηση. Ο εισηγητής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις δηλώσεις σας Θα ήθελα να στηρίξω και την αντιμετώπιση που έχει για το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τις ίδιες ανησυχίες εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα της συνολικής αντιμετώπισης της, των, της, προσωπικής, της προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων, γιατί είναι κάτι το οποίο απτέται και ε, του εσωτερικού συστήματος του δικού μας, για τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι δηλαδή προσπαθούμε να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και πως όταν ακούω τις δηλώσεις ιδιαίτερα της Ευρωπόλ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικά αυτά που λέτε η Ευρώπη έχει συνηθίσει ουσιαστικά να συνεργάζεται ε, με τις υπόλοιπες χώρες ε, με τις χώρες μέλη και να μεταφέρει στις χώρες μέλη πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται η Ευρωπόλ. Και όταν μιλάμε για διμερείς συμφωνίες, η μετατροπή υπάρχουσών συμφωνιών σε ένα νέο πλαίσιο είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται η Ευρωπόλ με τα διάφορα κράτη-μέλη. και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε ποιες είναι οι υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες. Όταν ακούω σαν παράδειγμα ότι υπάρχουν πολλαπλές απόψεις για το ποιες είναι οι συμφωνίες αυτές, διαρωτώ με αν η Ευρωπόλ γνωρίζει όλες αυτές τις διμερείς συμφωνίες και τα επίπεδα προστασίας τα οποία εφαρμόζονται. Νομίζω ότι δεν γνωρίζετε ακριβώς το ποιες είναι και πόσες και γι' αυτό είναι συμφέρος των κρατών μελών να ρυθμίσουν το συγκεκριμένο θέμα στο εσωτερικό της Ένωσης. Όταν αναφέρεται κανείς στις ε, αρχές επιβολής τάξεως που λειτουργούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γνωρίζουν τι συμφωνίες είναι σε ισχύ και θα πρέπει και το Eurojust να είναι ενήμερο για το υπάρχον πλαίσιο και για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με τα κράτη-μέλη και με τις κυβερνήσεις. Ίσως αυτή θα είναι η συζήτηση που θα πρέπει να γίνει. Οι δύο συνάδελφοι θέλουν ήδη το λόγο και ο κύριος Μέλντερ και ο κύριος Πρόντς η συμφωνία βασίζεται στην προϋπόθεση ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές, αλλά η συμφωνία θα υπογραφεί όχι εξ του Κογκρέσου, αλλά της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Όταν ξέρει κανείς τι ισχύει συνταγματικά ε, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα η κυβέρνηση να δώσει εγγυήσει για τη συμβατότητα των αποφασεών της με το Σύνταγμα. Οπότε τι ακριβώς ε, μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Ένωση έτσι ώστε οι αλλαγές αυτές πράγματι να υπάρξουν. Ας συλλέξουμε πρώτα όλες τις ερωτήσεις και μετά οι πανελίστες θα πάρουν το λόγο να απαντήσουν. Εγώ στην ουσία θα ήθελα να ακούσω τον τελευταίο μιλητή ε, λίγο περισσότερο γιατί πολύ μου άρεσαν αυτά τα οποία είπε. Υπάρχει το θέμα του επίπεδου προστασίας το οποίο ε, έχει από τον Σεπτέμβριο του 2001 ε, ε, έχει χαμηλώσει σε πάρα πολύ, ε, σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Έχουν γίνει τέτοιες προτάσεις και για τις θέως κομμουνιστικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάρα πολλές διαφορές όμως σε σχέση με τα επίπεδα προστασίας, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου. και η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Στη δική μου χώρα την Ουγγαρία μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουν γίνει κάποιες πρώτες προσπάθειες από τη νέα κυβέρνηση, τη συντηρητική κυβέρνηση να ξεκινήσουν με μια νέα υπηρεσία α, αντιτρομοκρατική, ιδιαίτερα ακριβή και ισχυρή είναι κάτι το εντελώς νέο με πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που σίγουρα είναι τόσο ισχυρή υπηρεσία που θα βρει τους τρομοκράτες. Κάποιες τέτοιες τάσεις υπάρχουν, πρέπει να δείξουμε κατανόηση. Εσείς σαν πανεπιστημιακός έχετε διαπιστώσει τέτοιου είδους τάσεις και αλλαγές στις διάφορες τεοσκομμουνιστικές χώρες. Μούλντερ. Η Γερμανία αρνήθηκε μια συμφωνία πρόσφατα επειδή δεν υπήρχαν αρκετές εγγύσεις. Θεωρήθηκαν ανεπαρκείς από την Bundesbank. Ξέρουμε ακριβώς ποια κρατημέλη έχουν συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά πόσο αυτές οι συμφωνίες είναι δημόσιες, κατά πόσες έχουν επικυρωθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά αυτό το θέμα. Η Europol, η Eurojust κάνουν κάτι ώστε να ξέρουμε περισσότερα. Σε αυτό το τελευταίο θα σας απαντήσω εγώ, γιατί ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό και συζητήσαμε στην Ολομέλεια και η Επιτροπή τι μας είπε, δεν ξέρουμε τίποτα. Μερικές φορές βρίσκουμε κάποια πραγματάκια, κάποια χαρτιά που έχουν πέσει από το φωτοτυπικό για παράδειγμα και έτσι λιγάκι παίρνουμε μια ιδέα για το ποια χώρα έχει κάνει τι. Ελάχιστα πράγματα όμως ξέρουμε. Για τη Γερμανία ξέρουμε λοιπόν ότι με ανοιχτό τρόπο, με διαφάνεια έχει κάποια συμφωνία η Αυστρία και η Γερμανία, τα μέσα ενημέρωσης δηλαδή, τα έχουν αναφέρει και έχει γίνει συζήτηση στην Bundesbank λοιπόν. Από μας η κυβέρνηση αρνήθηκε ότι υπήρξαν συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, μετά ε, άρχισαν να λένε ναι, ναι, αλλά διαπραγματευόμαστε ακόμα. Η ουσία είναι ότι δεν ξέρουμε. Στη δημοκρατική Ευρώπη δεν ξέρουμε. Είναι ζωτική σημασία όμω να μάθουμε. Θα ζητήσω λοιπόν από τους προσκεκλημένου μας να απαντήσουν, ξεκινώντα από τον κύριο Κόρφ, με την αντίθετη σειρά δηλαδή. Για διεθνεί συμφωνίες. Κοιτάξτε, πολλά έχουν γίνει για να είναι δεσμευτικές αυτές οι συμφωνίες. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια διαφορά για το αν είναι δεσμευτικές διεθνώς κάποιες συμφωνίες, είναι σε εθνικό επίπεδο. Εδώ εξαρτώμαστε από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τους εθνικούς. Από πλευράς Αμερικής δεν έχω τίποτα που να δείχνει ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και εκεί. Ότι δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους κανόνες ένας Ευρωπαίος πολίτης στα δικαστήρια στις ΗΠΑ. Πολύ καλά αυτά που λέτε. Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινούσα αλλιώς με κριτική στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική, αλλά με πρόλαβε ο πρέσβης. Έχω μαζί μου ένα βιβλίο. Αυτό. Της δεκαετία του 70. Είπατε είμαι ακαδημαϊκός, ναι. Αλλά είμαι και ακτιβιστής στα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεργάζομαι με τη Διεθνή Αμνηστία. Κοιτάξτε, τι έχει γίνει στη Γερμανία και όχι μόνο, στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες και στον Ηνωμένο Βασίλειο με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε από τη μια την ιδεολογική μάχη για την ασφάλεια και τις δράσεις της αστυνομίας όσον αφορά κάποιες εγκληματικές ε, πράξεις. Η τάση είναι επικίνδυνη. Η αστυνομία και το βλέπετε αυτό στις διάφορες συμφωνίες. Πρέπει να υπάρχει πραγματική ένδειξη ότι ένα άτομο εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στο τρομοκρατικό περιβάλλον. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε ο Σεμπάστιαν είναι ακριβώς τι σημαίνει εγκληματική δραστηριότητα, ότι επεκτείνουμε αυτή την έννοια. Ακούσαμε τρομοκρατία, επεδεραστία, είναι δύο ξεκάθαρα εγκλήματα. Εντάξει, βέβαια είναι τρομοκρατική ενέργεια να βάζει μια βόμβα και να σκοτώνεται κόσμος. Όμως πώς εμπλέκεται κανείς έμεσα ή άμεσα σε ένα τρομοκρατικό περιβάλλον. Ένας Γερμανός που έχει ζήσει τη δεκαετία του 70, δεν ξέρω, ο κύριος Άλμπρεχτ βέβαια είναι πιο νέος, αλλά για τον Μπούκεναχάου διάφοροι ακαδημαϊκοί διώχθηκαν τότε επειδή παραδημοσίευσαν άρθρο ανώνυμο και κάποιος άλλος σκέφτηκε ότι αυτό είναι στήριξη στην τρομοκρατία. Άρα λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καταπολέμηση εγκλημάτων που έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι τελικά όμως υποστηρίζουν κάτι άλλο. Κάποιος που γράφει ένα φυλάδιο όπου υποστηρίζει τη Χαμάς. Μπορεί να είναι τρομοκρατικό έγκλημα στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά βάσει της νομοθεσίας στη Γερμανία στην 89-98 που μιλάει για στήριξη στην τρομοκρατία μπορεί να είναι ηθική στήριξη. Δηλαδή υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη και πιέσεις που μας έρχονται από το Συμβούλιο και από τις κυβερνήσεις να μπουν σε αυτές τις συμφωνίες τα πάντα. Μα είναι πολύ επικίνδυνο. Με ανταλλαγές ονομάτων. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πει «Α, ή δαχτυλικό, το δαχτυλικό αποτύπωμα, ότι αυτό μοιάζει με κάποιον που έχουμε εμείς». Τελικά τι, η συμμετοχή σε μια διαδήλωση, το να έχει ρίξει κανείς μια πέτρα σε μια διαδήλωση, είναι τρομοκρατία για ορισμένε χώρε, αν πρόκειται για πολιτική διαδήλωση. Δηλαδή, οι κίνδυνοι δεν έχουν τέλο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο αυτά. Ευχαριστούμε. Τώρα, ο κύριος Σάιν. Ευχαριστώ. ετέθηκε ένα ερώτημα ως προς την κατάσταση στη Γερμανία και σε ποιο βαθμό η Γερμανία έχει απορρίψει αυτή τη μερή συμφωνία. Δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Η συμφωνία πρέπει να περάσει από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα, δηλαδή την Bundestag και την Bundesrat και εγκρίθηκε, αλλά λόγω τη ιδιαίτερη κατάσταση και τη ομοσπονδιακή δομή τη Γερμανία ε, υπήρξε ανάγκη για κάποιες διατυπώσεις οι οποίες ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί έτσι ώστε να θεωρηθεί περαιωμένη η κύρωση. Αυτό οφείλεται στις ε, ελλείψεις, στα κενά αυτής της συμφωνίας που σας σήμερα νωρίτερα. Νομίζω ότι μπορούμε κατά τα άλλα να επισημάνουμε μέσα από τις κοινέ αυτές δηλώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν τα, τις ελλείψεις αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, ε, πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μια νέα συμφωνία. Η υπηρεσία μας θεωρεί πολύ σημαντικό να θεμελιωθούν για τον ε, θυγόμενο δικαιώματα δυνάμει νέα νέας συμφωνίας που θα του επιτρέπει εφόσον κυρωθεί η συμφωνία και εφαρμοστεί και στις ΗΠΑ να προσφεύγει στα Αμερικανικά δικαστήρια. Εάν όμω αυτή η διαδικασία μετατραπεί σε μια διοικητική μόνο, που δεν δεσμεύει δηλαδή τα δικαστήρια των ΗΠΑ, τότε ουσιαστικά ε, απογυμνώνεται από την αξία και τη σημασία της μια τέτοια συμφωνία. Ευχαριστώ, κυρία Γκαμπρέλτσιτς. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ Eurojust και Ηνωμένων Πολιτειών ε, της Αμερικής, οι συμφωνίε όσο μας αφορούσαν ήταν οι εξή. Έγινε η διαπραγμάτευση έω προς το σχέδιο, επί του σχεδίου και όπως είπα και νωρίτερα πολύ προσοχή δόθηκε στις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων Εγκρίθηκε το σχέδιο από το Κοινό Εποπτικό Συμβούλιο, το Συλλογικό Όργανο της Eurojust και επιπλέον το Συμβούλιο και μόνο αφού πέρασε από αυτές τις τρεις διαδικασίες μπόρεσε να εγκριθεί η συμφωνία. Οι εσωτερικές διαδικασίες και των δύο πλευρών φυσικά ακολουθούν την εφαρμόσιμη νομοθεσία, την εφαρμόσιμη νομοθεσία, είτε είναι εθνική είτε είναι διεθνής. Επομένως, ε, όταν ε, ολοκληρωθούν ή όταν ολοκληρώθηκαν καλύτερα οι εσωτερικές διαδικασίες των δύο πλευρών, ε, θεωρήθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί και τίθεται σε ισχύ η συμφωνία με μια κοινοποίηση των πράξεων κύρωσης. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο, αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Όχι, δε, στρέφομαι προς συναδέλφους αν θεωρούν ότι δεν έχει απαντηθεί κάποια ερώτησή τους. Μάλλον είναι ικανοποιημένο. Κύριο Σέρτινγκ, ευχαριστώ και εγώ θα είμαι σύντομος. Η συμφωνία μας ε, ακολουθεί λίγο πολύ αυτό που συνέβη και με τη Eurojust. Ε, ανταλλάξαμε όλες τις πληροφορίες μας. Ε, είχαμε και συμφωνίες με τα κράτη-μέλη. Ανεξαρτήτως του με ποια χώρα είχαμε την σύμπραξη αυτή, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία. Κατά τα άλλα, διμερεί συμφωνίε ε, δεν είναι πάντοτε γνωστέ. Άλλε είναι κοινέ στη σπάση, άλλε έχουν ε, απόρριτα παραρτήματα. Ίσως θα είναι καλό να υπάρχει σχετική ενημέρωση. Απόφαση δική σα, βέβαια, αλλά ίσως θα πρέπει να το χειριστεί και η Επιτροπή. Η Πρόεδρος. Μα η Επιτροπή έχει επεκτηθεί ασδήποτε ευθύνε στην υπόθεση αυτή. Ασφαλώ όμως θα μα ε, απασχολήσει και πάλι το θέμα. Ο κύριο Σιγητή έχει να πει κάτι ακόμη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Νομίζω ότι υπογραμμίσαμε, περιγράψαμε μια σειρά από ζητήματα που ενδιαφέρουν και την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο βεβαίω δεν έχει φτάσει ακόμη στην ολοκλήρωση διαδικασία για την έγκριση τη ε, προτινόμενη εντολή, αλλά ασφαλώ θα διατυπώσουμε τι θέσει μα, απερίφραστα. Και όταν δούμε και πώς εξελίσσονται οι ε, διμερείς αυτές ε, διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις για μια συμφωνία πλαίσιο που τελευταία ανάλυση πρέπει να αποτελεί και σημείο αναφοράς γιατί αποτελεί μια κοινή βάση πάνω στην οποία συνάπτουμε τις διμερείς μας συμφωνίες. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερως που βλέπω ε, οργανώσει υπηρεσίες όπως η Europol και η Eurojust που μας στηρίζουν σε αυτό μας το μέλημα και χαίρομαι διότι το αίτημα δεν έχει να κάνει μόνο με τα ε, πολιτικά δικαιώματα, αν και πάνω από όλα αφορά τα πολιτικά δικαιώματα, αλλά και την ε, ανάγκη για τις δημόσιες αρχές, για τις κρατικές αρχές, τις ευρωπαϊκές, να έχουν ε, καλό επίπεδο και νομικής ασφάλειας και ύψιστη η προστασία των δικαιωμάτων. Αυτό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έξω από αυτήν στη σχέση μας με τους εταίρους, με τις άλλες χώρες. Τώρα θα δούμε πώς το ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας αυτής θα αντιμετωπιστεί από το Συμβούλιο. Ελπίζω να μας ακολουθήσει, γιατί είναι για μας κρίσιμη σημασία σε μια τέτοια συμφωνία να μην υπάρχει μερολεπτική προσέγγιση. Γιατί αυτό βέβαια θα επηρεάσει κάθε νέα συμφωνία. Εμείς εκπροσωπούμε τον Ευρωπαίο πολίτη. Ο Ευρωπαίο πολίτης θέλει να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του και στη τελευταία ανάλυση θέλει και να ε, βεβαιώνεται ότι μπορεί να επιβάλλει το σεβασμό των δικαιωμάτων του. Εάν το εξασφαλίσουμε εμείς αυτό, τότε θα έχουμε κάνει τη δουλειά μας ως βουλευτές. Γι' αυτό και Ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε στον δρόμο αυτό μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τους παρόντες εδώ, τους χιώδει ηγητέ δηλαδή, αλλά και εμένα ως εισηγητή που έχω αναλάβει το θέμα αυτό. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Δεν μπορώ παρά να πω κι εγώ, καταλήγοντας, ότι ελπίζω πως ε, το Συμβούλιο ως συνομοθέτης θα φροντίσει να οργανώσει αντίστοιχες ε, με τη δική μας ακρόαση ώστε να ενημερωθεί και εκείνο για τις ανησυχίες και τα ε, διλήμματα που προκύπτουν ε, από αυτό το θέμα. Στο παρελθόν ξέρουμε ότι δεν το έπραξε και ξέρουμε ότι δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένο. Εμείς πάντως έχουμε μάλλον ε, την αντίθετη παράδοση. Πάντοτε ενημερωνόμαστε από τους προσκεκλημένους μας και στηρίζουμε τις αποφάσεις μας στις δικές τους γνώσεις και την πείρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια ολόκληρης συνεδρίασης. Τελειώνουμε εδώ και ξεκινάμε σε πέντε λεπτά τη συνεδρία των συντονιστών για τους παρόντες. Και ευχαριστώ τους διεμένες, λέει πρόεδρος. Ευχαριστούμε.